Colleagues, please, can we start our meeting? Παρακαλώ, να αρχίσουμε. Πρώτο θέμα έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Να θεωρήσουμε ότι είναι κρίθη. Ευχαριστώ. Να εγκρίνουμε και τα πρακτικά της συνεδρίασης ε, της 12ης Μαρτίου. Υπάρχουν παρατηρήσεις, όχι, ευχαριστώ. Λοιπόν, να περάσουμε στη συζήτηση για τις τρομπολογίες στην έκθεση Μπούλμαν Φερνάντες. Πολύ σημαντική συζήτηση που θα διεξαγάγουμε. Λάβαμε 1396 τροπολογίες. Βέβαια μεγάλος αριθμός, αλλά λόγω της σημασίας του θέματος αναμενόμενος. Να σχολιάσω προσωπικά. Είναι προφανές ότι είναι διαφορετικές αυτές οι τροπολογίες, αλλά διαπιστώνω μια κάποια σύγκληση. Μια συγκλίνουσα προσπάθεια των μελών του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής να έχουμε ένα πρόγραμμα αποδοτικό που να εγγυάται τη συμπληρωματικότητα των επενδύσεων και να έχει και δημοκρατικό έλεγχο. Καλή βάση για την εργασία μας για να προετοιμάσουμε την ψηφοφορία που θα πρέπει να γίνει σε λιγότερο από ένα μήνα και έχουμε και τη σημαντική γνωμοδότηση που θα λάβουμε στις 14 Απριλίου αλλά είμαι σίγουρος ότι οι εισηγητές θα προετοιμάσουν την εργασία με βάση και το κείμενο και τις συζητήσεις. Ένα καλό κείμενο λοιπόν πιστεύω ότι θα έχουμε για να αρχίσουμε τη διαπραγματεύση με το Συμβούλιο. Ζάων, θέλεις να προσθέσεις? Ναι βεβαίως, ε, χαιρετίζω τις τροπολογίες από τους ε, δύο εισηγητές και όλους τους συναδέλφους. Χαίρομαι για το πόσο ενεργή ήταν η συμμετοχή όλων αυτό καταδεικνύει ότι μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Πρέπει λοιπόν να καταλήξουμε στους σωστούς συμβιβασμού για να έχουμε ένα κείμενο υψηλής ποιότητας που μέσα στα περιορισμένα χρονικά περιθώρια να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας ούτω ώστε να προσδώσει στην Ευρώπη αυτήν την επιπλέον δυναμική για να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας μέσω επενδύσεων. Ρομπέρτο, παρακαλώ, προεδρεύστε περαιτέρω. Ευχαριστώ Ζω. Ποιος θα ξεκινήσει, ο Ιωνάς. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ο Ιωνάς Φερνάνδας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον εισηγητή Μπούλμαν, τον συνεισηγητή μου για όλη την εργασία που έχει καταφέρει και τους σκιώδεις για τη συνεργασία μας. Έχουν με λοιπόν πολλές τροπολογίες, ιδίως τη Ήτρα και τη Τραν, πράγμα που σημαίνει ότι οι ευρωβουλευτές ε, συνεργάστηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό και δείχνει επίσης τη σημασία που δίνουν σε αυτό το θέμα γιατί το ταμείο αυτό είναι σημαντικό για τις επενδύσεις <coughs> για την εμπάθυνση της ενιαίας αγοράς αλλά και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα επιτρέψει αύξηση της απασχόλησης, ανάπτυξη και θέλει να είναι η έκφραση, η ανταπόκριση σε επανειλημμένες εκκλήσεις του Κοινοβουλίου ώστε πέρα και από αυτό το ίδιο το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων να συμμετάσχουν και τα διαρθρωτικά ταμεία και να υποφεληθούν από τα οποία υποφελούνται ήδη, τα κράτη-μέλη. Πράγματι, οι τροπολογίες έχουν κοινά στοιχεία, δηλαδή να δημιουργηθεί, ζητούν να δημιουργηθεί ένα ταμείο ένα σχέδιο μάλλον επενδύσεων το οποίο πρώτο προτάθηκε τον Ιούνιο το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές αλλά ίσως δεν δώσαμε αρκετό χρόνο σε αυτές τις συζητήσεις και είδαμε και πόσο ποιοτικέ είναι οι τροπολογίες Άρα πρέπει όντως να καταλήξουμε σε συμβατικές τροπολογίες. Πρέπει να καταλήξουμε σε συμβατικές τροπολογίες, οι οποίες δεν θα πρέπει να θέτουν ένα αμφιβόλο τη συνοχή του κανονισμού αυτού. Αυτό, αυτό που επιδιώκουμε είναι η διαδικασία αυτή να καταλήξει επιτυχώς. Όλες οι προσπάθειες που έγιναν για τη χρηματοδότηση έχουν ένα κοινό στόχο, ο οποίος είναι να μειωθεί η επίπτωση που έχει αυτό το πρόγραμμα Λοιπόν, λοιπόν, έχουμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Ελπίζω να έχουν επιληθεί τώρα. Έλεγα λοιπόν, η χρηματοδότηση Έλεγα λοιπόν, υπάρχει μια κοινή γραμμή για τη χρηματοδότηση. Θέλουμε να μειώσουμε στο μέτρο το δυνατό τις περικοπές στο συνδέοντας την Ευρώπη και την ορίζοντα 2020. Η πρότασή μας είναι να υπάρχει η αναγκαία ευελιξία για την ε, πρικοδότηση αυτού του ταμείου και πάνω από όλα θέλουμε αυτή η η χρηματοδότηση να μην έχει καμία επιπλέον προϋπόθεση, καμία επιπλέον αρεσιμότητα πέραν της εγγύησης. Κανείς να μην... Τι να κάνω, να μιλήσω γαλλικά, γιατί δεν μοιάζει να λειτουργεί η διερμηνία. Καλά, καλά. Να επιχειρήσω άλλη μια φορά, πώς έλεγα λοιπόν. Υπάρχει μια κοινή γραμμή για τη χρηματοδότηση. Θέλουμε να μειώσουμε την επίπτωση που έχει στον ορίζοντα 2020 και στο μέσο συνδέοντα την Ευρώπη. Αυτή η κοινή γραμμή μας βρίσκει όλους σύμφωνους. Θέλουμε ευελιξία λοιπόν, χωρίς να διακυβεύεται η αξιοπιστία. Θέλουμε να ενισχύσουμε το πρόγραμμα αυτό. Κανείς δεν αφισβητεί τα 16 δις εγγύσεων. Αυτό που προσθέτουμε είναι ότι αυτά τα 16 δις πρέπει να διατηρηθούν. Αυτό τονίζουμε, χωρίς άλλε συνθήκες και προποθέσει. Όχι, λειτουργεί η γερμανική μετάφραση, λέει ο πρόεδρος. Αλλά να μην μιλάτε παρακαλώ. Also die Übersetzung ist miserabel, wird ständig und Διαρκώς διακόπτεται η διερμηνία προς τα γερμανικά, λέει ο πρόεδρος. sorry, I'm not the condition to judge the quality of the German translation. Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να κρίνω την ποιότητα της ε, ε, γερμανικής διερμηνίας. Υπάρχει διερμηνία. Αν αφήσετε τους διερμηνείς να εργαστούν, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Λοιπόν, θα επιχειρήσω να ε, ολοκληρώσω την ε, διερμηνία μου στα πορτογαλικά. Όπως έλεγα λοιπόν, θέλουμε ένα αξιόπιστο πρόγραμμα. Αυτό είναι η προϋπόθεση για να επιτύχει θέλουμε να έχει το μέγιστο αξιοπιστίας και λέγαμε ότι αυτή η εγγύηση πρέπει να είναι χωρίς προποθέσει, να είναι οριστική, αμετάκλητη. Κανείς να μην μπορεί να την αμφισβητήσει αυτές ε, τις εγγύσει που θα δώσουν τα 16 δι. Θέλουμε να μειώσουμε, όπως έλεγα επίση, την επίπτωση στο συνδέοντα στην Ευρώπη και τον ορίζοντα 2020. Γι' αυτό πέρα από τι προτάσει που κάναμε, στα πλαίσια του πλεονάσματος που μπορεί να προκύψουν από τη χρήση αυτού του ταμείου και λέμε ότι αν υπάρξει πλεόνασμα θα πρέπει να επιστρέψει στις δύο προηγούμενες χρηματοδοτήσεις. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει ισχυρή δέσμευση και από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή ότι στα πλαίσια της αναθεώρησης ε, το 17 ε, των δημοσιονομικών προοπτικών θα επιχειρήσουμε να έχουμε την ε, απόλυτη δέσμευση ή την όσο το δυνατόν πιο ισχυρή δέσμευση ότι τα προγράμματα και οι γραμμές που αξιοποιήθηκαν για να δημιουργηθούν αυτές οι εγγυήσεις να μπορούν να αποκατασταθούν στα πλαίσια ακριβώς αυτής της αναθεώρησης το 17 Θέλουμε λοιπόν η αναθεώρηση του 17 να μας βοηθήσει να αποκαταστήσουμε τις γραμμές που, που ε, περιεκόπησαν για να δημιουργηθεί αυτό το Ταμείο Εγγύσεων. Έχει γίνει μια άλλη πρόταση για να πρικοδοτηθεί το Ταμείο αυτό. Τα πρώτα χρόνια δεν υπάρχει περιθώριο απολειών, δηλαδή από αυτά τα 8 δις του Ταμείου Εγγύσεων Ε, να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες. Θέλουμε το επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο να διατηρήσει αυτή τη δυνατότητα. Αλλά στο μέτρο που θα χρειαστεί. Δηλαδή, αν δεν χρειάζεται να είναι τόσο μεγάλη η χρηματοδότησή του, να το δούμε. Νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή πρόταση για να επιτύχουμε αυτό το στόχο της μη μείωσης τελικά του ορίζοντα 2020 ε, και του μέσου συνδέοντα την Ευρώπη. Για τα άλλα θέματα, συγκεκριμένα όλα όσα αφαιρούν τη διακυβέρνηση του Ταμείου, την επιλογή προγραμμάτων, την ε, σύσταση του Διοικητικού Συμβουλίου, Βεβαίως θα κάνουμε πρόταση, αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να μην υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις. Κάναμε μια πρόταση τροπολογίας όπου λέμε ότι αυτή η Διοικητική Επιτροπή δεν θα πρέπει να περιέχει εκπροσώπηση των κρατών μελών για να μην υπάρξει πολιτικοποίηση τη λειτουργία του. Έχουμε και διάφορε τροπολογίε για τι κατεξοδότηση πράξη. Να έχουμε υπόψη μα ότι είναι σημαντικέ για το Κοινοβούλιο αυτέ, αλλά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να ξαναξεκινάει διαρκώ και να επαναλαμβάνεται η συζήτηση επιθεμάτων ήδη αποφασιστέντων. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Πρέπει να δούμε πώ θα επιλέξουμε τα προγράμματα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να είναι περίπλοκη η διαδικασία επιλογής αν συμπεριλάβουμε υπερβολικά πολλά κριτήρια για την επιλογή των προγραμμάτων, ε, αν λέμε ότι πρέπει να υπάρχει υψηλή προστιθέμενη αξία για την απασχόληση, την ποιότητα κτλ, στο τέλος θα αποκλείσουμε προγράμματα που μπορεί και να είναι σημαντικά. Αλλά το πιο σημαντικό, όπως είπα λοιπόν, είναι η αρχή της προσθετικότητας. Επίσης, να ε, επιδιώκουν μία ε, ανάπτυξη ε, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη και να ε, τηρούν φυσικά και τις τεχνικές προϋποθέσεις. Νομίζω ότι μπορούμε τον Ιούνιο να έχουμε ένα αξιόπιστο τέτοιο ταμείο, αλλά για να γίνει αυτό δεν θα πρέπει να ξανανοίξουμε ή να ανοίγουμε συνέχεια τη συζήτηση για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Η Ευρώπη χρειάζεται μια τέτοια ε, δράση, ένα τέτοιο εγχείρημα. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους. Νομίζω θα τα επιτύχουμε και να ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα τον κύριο Μπούλμαν με τον οποίο συνεργάστηκα πάρα πολύ και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μπούλμαν τώρα. Κύριε Πρόεδρε, η συνδυασμένη εργασία των επιτροπών μας, αγαπητοί συνάδελφοι, και συγκεκριμένα του Χωζέ Μανουέλ, τόνισε ότι η εργασία αυτή έγινε από όλους μας μαζί, όλους τους συναδέλφους. Υποβλήθηκαν, λέει ο συγητής, γύρω στις 2.000 τροπολογίες. Αυτό νομίζουμε ότι είναι ένδειξη του ενδιαφέροντος που υπάρχει. Ευχαριστούμε τους συναδέλφους για το πόσο τους ενδιαφέρει τόσο πολύ και πράγματι, πράγματι το θέμα το αξίζει. Είναι μια συμβολή στον δημοκρατικό πολιτισμό και στην δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης και δημοκρατίας. Αυτή η πλατιά συμμετοχή των συναδέλφων. Και γι' αυτό είναι και τόσο υψηλή η πίεση. Πίεση να καταλήξουμε σε ένα υψηλής ποιότητας κείμενο, τηρώντας επίσης τις προθεσμίες τις οποίες ανέφερε ο Ζωζέ Να κάνω λοιπόν μία παρατήρηση εισαγωγικά. Θα επιτύχουμε αυτόν τον σημαντικό στόχο μόνο αν υπάρξει καλή συνεργασία αν διατηρήσουμε ε, αυτήν την ε, καλή πρόθεση να επιτύχουμε συμβιβασμούς πέρα από επιτροπές, πέρα από πολιτικές ομάδες και ευχαριστώ πάρα πολύ που υπάρχει αυτή η καλή πρόθεση γιατί το αξίζει το θέμα. Ξέρουμε πόσο έντονη είναι η εργασία για τους συνεργάτες μας ε, και πολλούς που μας βοηθούν που δεν τους ε, βλέπουμε κάθε μέρα τις μεταφραστικές υπηρεσίες για παράδειγμα και τους συναδέλφους που εδώ μας παρέχουν τη διερμηνία και ξέρω ότι η πίεση για όλους μας είναι πολύ υψηλή θέλω εκπεφρασμένα να ευχαριστήσω όλες τις καμπίνες της διερμηνίας για την ε, πολύ καλής ποιότητας εργασία τους Ξέρω πως έτσι το βλέπει και ο συνάδελφος Βέρνερ Λάγγεν. Γι' αυτό νομίζω ότι μπορώ να μιλήσω και από πλευράς του. Τώρα, επί της ουσίας. Να επιχειρήσω. Να αναφέρω όλα τα επιχειρήματα κατά τομής. Ένα σημαντικό τομέας, τον οποίο πρέπει να συζητήσουμε, είναι με ποιο, με ποιο τρόπο θα κάνουμε τις ε, διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο. Βλέποντας τις τροπολογίες των συναδέλφων, διαπιστώνω ότι γενικά στηρίζεται η γραμμή των εισηγητών, υπάρχουν διαφοροποιήσεις, υπάρχουν συνάδελφοι που είναι πιο φιλόδοξοι, λέγοντας ότι το Εύση θα πρέπει να έχει τη δική του νομική προσωπικότητα. Ενδιαφέρουσα πρόταση, γιατί νομίζω ότι αφορά και το μέλλον. Θα μπορούσε να μας βοηθήσει πολύ στο μέλλον, αλλά τώρα επειδή είναι τόσο λίγος ο χρόνος, εάν θα το καταφέρουμε, αλλά είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε μεταξύ των σκιώδων εισηγητών και εισηγητών. Μια σημαντική πρόταση είναι αυτή λοιπόν από την πλευρά του ΕΛΚ. Η πρόταση λοιπόν αυτή λέει να υπάρχει ένα εποπτικό συμβούλιο όπου όλες οι τράπεζες και όλοι οι μεσάζοντες που θα εργάζονται με αυτές τις ε, εγγυήσει της Ένωσης που παίζουν λοιπόν μεγάλο ρόλο και πρέπει να συνεργαστούν στενά βλέπω ότι αυτό, αυτή την πρόταση υπάρχει ευρεία υποστήριξη. Επόμενο θέμα πώς θα διασφαλίσουμε την επαρκή πρικοδότηση του Ταμείου. Ορισμένοι συνάδελφοι εκφράζουν ε, την απογοήτευσή τους για το ότι ορισμένα κράτη-μέλη δεν είναι διατεθειμένα ή δεν είναι σε θέση να συμμετάσχουν στη χρηματοδότηση. Νομίζω όμως ότι πρέπει να χαιρετήσουμε το γεγονός ότι είπαν πολλοί ότι θα συμμετάσχουν μέσω εθνικών οργανισμών προώθησης επενδύσεων στην ε, χρηματοδότηση των προγραμμάτων επιμέρους. Όλη λοιπόν η λειτουργία του ΕΦΣΙ θα βοηθηθεί μέσω αυτών των εθνικών και περιφερειακών συμβολών. Και εδώ βλέπω να υπάρχει ευρεία συνένεση. Βλέπω τις τροπολογίες των φιλελεύθερων να αναφέρουν, όπως είπε ο Ραμόν, ότι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τις περιφέρειες. Οι περιφέρειες παίζουν μεγάλο ρόλο στην ε, εξέβρεση των πιο προσαρμοσμένων λύσεων για να βοηθήσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή για να βελτιώσουμε τις υποδομές και να αντιμετωπίσουμε τις ελλείψεις στον τομέα των υποδομών. Και εδώ βλέπω ευλία, ευρεία πλειοψηφία. Οπότε τίθεται το ερώτημα ε, ποιο θα είναι το αρχιεκτονικό σχέδιο αυτού του νέου κτηρίου και συγκεκριμένα ε, αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Επενδύσεων. Επ' αυτών υπάρχουν διαφορετικές ε, αντιλήψεις για το πώς περαιτέρω θα διαμορφωθούν. Έχουμε προτάσεις από το ΕΛΚ, από τους σοσιαλιστές, από τους πράσινους, από την ΚΟΕ, οι οποίοι μας λένε ότι αυτή, αυτό το Διοικητικό Συμβούλιο, Steering Board Committee, πρέπει να ενισχυθεί και το EFDD. Αλλά οι φίλοι από τους συντηρητικούς λένε ότι ότι το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να καταργηθεί. Γιατί η ίδια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχει τις κατάλληλες δομές. Άρα πρέπει να το συζητήσουμε. Δεν είναι δυνατόν από τη μία να ενισχύσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο και από την άλλη να το καταργήσουμε. Πρέπει να αποφασίσουμε τη γραμμή μας από αυτού. Εγώ, ε, εκτός αν με πείσετε για κάτι διαφορετικό, δεν θεωρώ ότι μπορούμε να το καταργήσουμε γιατί εκεί θα συμμετάσχουν και όλοι οι μέτοχοι. Αυτοί που θα πρέπει να εκτελέσουν τις αρμοδιότητες που θα τους χορηγήσουμε. Δηλαδή θα συμμετάσχει και η Επιτροπή και η Τράπεζα Επενδύσεων. Σε πολλές συζητήσεις έπαιξε ρόλο μία αμφιβολία. Όπως συχνά πώς θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω αυτό το ταμείο, πόσο ανοιχτό θα είναι προς τρίτους. Γιατί ορισμένοι θεωρούν ότι όποιος χρηματοδοτεί θα πρέπει να έχει λόγο και για την ε, απόφαση των επενδύσεων, τον προσανατολισμό των επενδύσεων, το προφίλ των επενδύσεων. Ορισμένοι λένε ότι εφόσον θα υπάρχει ιδιωτικό κεφάλαιο και μάλιστα εκτός της Ένωσης, ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή του χαρακτήρα του Ταμείου. Γι' αυτό το ΕΛΚΑ έχει καλές προτάσεις, οι οποίες μας προτείνουν ένα διαχωρισμό μεταξύ αυτών που λένε εφόσον πληρώνουμε θέλουμε να συμμετέχουμε και στη λήψη των αποφάσεων, αλλά οι συνάδελφοι κάνουν προτάσεις που λένε ότι δεν πρέπει να μπορούν άμεσα να συμμετάσχουν ακριβώς στην κατεύθυνση των χρηματοδοτήσεων του Ταμείου. Για την Επιτροπή Επενδύσεων τώρα. Και εδώ υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις. Ποια θα πρέπει να είναι η σύνθεσή της. Πολλοί συνάδελφοι λένε, όπως ε, ο κύριος Ζάντερ λέει, ότι πρέπει να είναι ανεξάρτητη η κυρία Γκρέσλε υπέβαλε τροπολογίες ότι πρέπει να συνδέεται με το κοινό συμφέρον και λέει ότι πρέπει ε, οι ισολογισμοί να είναι διαφανής να βλέπουμε πώς λειτουργεί το Ταμείο, οι πράσινοι ε, συνάδελφοι και άλλοι από το ΕΛΚΑ και οι σοσιαλιστές τονίζουν ότι πρέπει να εκπροσωπούνται Ευρέα συμφέροντα σε αυτήν την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Πώς θα δημιουργηθεί λοιπόν αυτή η Επιτροπή και συγκεκριμένα πώς θα οριστεί ο επικεφαλής της και ο αναπληρωτής του. Και επ' αυτού υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Η γενική τάση όμως του σώματος είναι σαφή. Δεν θα πρέπει να αγνοηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το καθορισμό των κατευθυντηρίων γραμμών και για τις αποφάσεις επί των, των κυρίων υπευθύνων. Δεν μπορεί να αγνοηθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί αυτό θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο για να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση από τον ενωσιακό προπολογισμό, Βέβαια τεχνικά πώ θα λειτουργήσει αυτό θα πρέπει να το διευκρινίσουμε. Οι λεπτομέρειε είναι ακόμη ανοιχτέ. Το αυτό ισχύει και για το θέμα πώς θέλουμε να συνοδεύσουμε τη λειτουργία του Ταμείου στο μέλλον. Θα πρέπει να πεθάνει από φυσικό θάνατο το Ταμείο ή θα πρέπει να του δώσουμε κάποια στιγμή τη δυνατότητα να μεταμορφωθεί. Υπάρχουν διαφορετικές τάσεις. Όμως η ευρεία συνένεση του σώματος είναι ότι μετά από τρία χρόνια πρέπει να κάνουμε μια επανεξέταση. Κανείς δεν λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε σε τρία χρόνια να σταματήσει Εάν έχει λειτουργήσει καλά, θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε περαιτέρω να το αναπτύξουμε. Με την κατάλληλη μορφή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τους δύο εισηγητές για τις παρουσιάσεις τους. Σας περάσουμε τώρα στους κοιόδης εισηγητές. Ο κύριος Κάρας το ο πρώτος ομιλητής. Κύριε Συμπρόεδρε, δεν νομίζω ότι τώρα ο κάθε σκιώδης θα πρέπει να επαναλάβει όλα όσα υπόθηκαν. Το αποφασιστικό είναι να προχωρήσουμε τη συζήτηση, να δούμε σε ποιους τομείς πρέπει να βελτιωθεί η έκθεση και σε ποιους ε, τομείς μπορούμε να συμφωνήσουμε. Υποστηρίζω λοιπόν αυτά που υπόθηκαν από τους δύο εισηγητές και στην ανάλυση τους. Έχουμε μια καλή βάση. Να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Σε πολλές εφημερίδες διαβάζω ότι ο αριθμός των τροπολογιών θεωρείται ως απόδειξη ότι το Κοινοβούλιο θέλει να μπλοκάρει αυτό το Ταμείο Εγγύσεων ή τουλάχιστον να κολλησιεργήσει. Πρέπει να είναι σαφές ότι μελετώντας ε, και το σχέδιο έκθεσης και τις τροπολογίες είναι σαφές ότι η ευρεία πλειοψηφία του σώματος επιθυμεί να λειτουργήσει αυτό το ταμείο. Θέλει να τηρήσει και τις προθεσμίες και θέλει απλώς να βελτιώσει σε τρεις αποφασιστικούς τομεί από πού θα προκύψει η χρηματοδότηση στη διακυβέρνηση και στη δυνατότητα δράση. ούτως ώστε να μην γίνει ένα ταμείο Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ΣΥΝ αλλά ένα Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων προσανατολισμένο προς το μέλλον ούτως ώστε να έχουμε ανάπτυξη και απασχόληση και για να γίνουμε παράγοντας στις παγκόσμιες επενδύσεις. Αυτό αυτός είναι ο στόχος μας. Και γι' αυτό λαμβάνει η χώρα μια δημοκρατική διαδικασία. Θέλω όμως να είμαι επίσης σαφής, σαφέστατος σε σχέση με το εξής. Όποιες τροπολογίες θέτουν εν κινδύνο αυτούς τους στόχους δεν θα μας βρουν σύμφωνους. Επίσης, κατά την ε, πολιτική μας ομάδα, κατά την πολιτική μου ομάδα, οι τροπολογίες πρέπει να έχουν δύο στόχους. Η χρηματοδότηση πρέπει να είναι σίγουρη και αμετάκλητη. Ναι ή όχι. Πρέπει να είναι λοιπόν ε, σαφές ότι πρέπει να ισχύουν αυτές οι δύο προϋποθέσεις. Γιατί αλλιώς δεν υπάρχει ασφάλεια επενδύσεων. Και αυτό θέτει εν κινδύνο την αναγκαία συμμετοχή ιδιωτικών επενδυτών. Αυτό το Ταμείο Εγγύσεων και οι στόχοι του μπορούν να λειτουργήσουν μόνο μέσω συνεργασίας ε, δημοσίων πόρων που θα είναι έναυσμα και η συμμετοχή των ε, ιδιωτικών επενδυτών που θα είναι το αποτέλεσμα του έναυσματος. Επίσης, οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται ανεξάρτητα. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ευνοιοκρατία και πολιτικές παρεμβάσεις. Γιατί αλλιώς οι ιδιωτικοί επενδυτές και τα ιδιωτικά προγράμματα δεν θα προκύψουν. Δεν πρόκειται περί αντιφάσεως. Ανεξάρτητες αποφάσεις και κοινοβουλευτική συμμετοχή. Δεν υπάρχει καμία πρόταση των εισηγητών που να είναι κατά αυτών των στόχων. Θέλουμε να υπάρχει σωστή διακυβέρνηση, αυτό θέλουν και οι εισηγητές, διότι θα υπάρξει και νοσιακή χρηματοδότηση. Και γι' αυτό η δομή διακυβέρνησης και η κατεξοδότηση πράξης δεν αντιφάσκουν σε σχέση με την ανεξάρτησία των αποφάσεων. Και κάτι ακόμη. στον τομέα της διακυβέρνησης. Στον τομέα των, ε, των, ε, των, των πλατφορμών της, των κλάδων και του προϋπολογισμού. Πρέπει να κάνουμε κάτι περισσότερο. Με βάση τις ε, προτάσεις και την ανάλυση που, έκανε, που έκαναν οι εισηγητές για να επιτύχουμε συμβασμούς που να ανταποκρίνονται τους στόχους και τις αρχές. Γι' αυτό καλώ όλους ε, να εργαστούν προς αυτή την κατεύθυνση με αυτόν τον τρόπο και προσβλέπω στην περαιτέρω συνεργασία. Thank you. Now... Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος Ευχαριστώ. Δεν θα επαναλάβουμε αυτό που είπαν οι συγητές. Τα έχουμε συζητήσει επανειλημμένα, συμμεριζόμεθα τη γραμμή εργασία τους και πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία για να στείλουμε μηνύματα και προς την κοινή γνώμη. Γιατί και εγώ, όπως και ο κύριος Κάρας, διάβασα ερμηνείες, κακόπιστες ή όχι, δεν ξέρω, που λένε ότι το Κοινοβούλιο θέλει να μπλοκάρει το Ταμείο. Δεν θέλει να προχωρήσει. Γιατί λένε ότι υποβάλαμε πολλές τροπολογίες. Το αντίθετο, οι 2.000 ε, τροπολογίες που έχουν υποβληθεί δείχνουν τι ενδιαφέρον υπάρχει εδώ στο Κοινοβούλιο για να προχωρήσει το Ταμείο. Αλλά από πλευρά του Κοινοβουλίου και από πλευρά Επιτροπή Προπολογισμών θεωρούμε ότι πρέπει να γίνουν ε, σοβαρέ βελτιώσει. Βελτιώσει του Ταμείου, τη αποτελεσματικότητά του και τη επίπτωσή του. Όσον αφορά την προσθετικότητα, αλλά και των επιπτώσεων που θα έχει για τον ενωσιακό προπολογισμό και γι' αυτό οι γραμμές που η σοσιαλιστική ομάδα προώθησε στο... για το θέμα αυτό είναι να μειωθεί η επίπτωση που θα έχει η δημιουργία του έψι στις γραμμές του προϋπολογισμού και μάλιστα τόσο σημαντικές όπως ορίζον 2020 και το μέσο συνδέοντας την Ευρώπη. Οι τροπολογίες λοιπόν που υποβάλαμε σε συμφωνία με τους συζητητές αλλά και ως σοσιαλιστική ομάδα από μόνοι μας στοχεύουν στη μείωση αυτής της επίπτωσης, αλλά οπωσδήποτε χωρίς να θέτουν κινδύνο το ταμείο, το επενδυτικό πρόγραμμα. Αυτό είναι το πρώτο μήνυμα που πρέπει να στείλουμε. Ό,τι κάνουμε είναι για να βελτιώσουμε και σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να διακυβευτεί αυτό το πρόγραμμα. Πρέπει να λειτουργήσει, το πιστεύουμε. Γιατί ε, θα είναι καλό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δύο κύριες καθευθυντήρες γραμμές από πλευρά σοσιαλιστών είναι πρώτον δεν θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο ούτε σωστό να αποφασίσουμε απριόρι για το από πού θα βγουν οι χρηματοδοτήσεις του ΕΦΣΥ. Πολύ πιο λογικό θα είναι να δουλεύουμε χρόνο το χρόνο έχοντας ε, πληροφόρηση για το πώς έχουν εκτελεστεί γραμμές του προπολογισμού και ποιες είναι ανάγκες του προγράμματος ούτω ώστε να έχουμε απεικόνηση του προπολογισμού καλύτερη και να δούμε από πού μπορούμε να βγάλουμε και πώς μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε λοιπόν την επίπτωση των προπολογισμών και το σαφές παράδειγμα γιατί αυτή είναι καλύτερη μέθοδος εργασίας είναι το 2015 τώρα το 2015 έχουμε την τύχη ότι το ίτερ δεν θα χρειαστεί 490 εκατομμύρια άρα υπάρχει χρήμα από εκεί για να το θέσουμε στο ΕΦΣΥ αν την απόφαση αυτή την είχαμε πάρει πριν από 4 μήνες δεν θα είχαμε καταλάβει ότι έχουμε χρήματα από το Ίτρε και θα πηγαίναμε αλλού να τα βρούμε. Αυτό μπορεί να συμβεί κάθε χρόνο. Γι' αυτό τι λέμε. Να δημιουργηθεί το Δαμείο Εγγύσεων. Αλλά χρόνο το χρόνο να βλέπουμε πώς θα το χρηματοδοτούμε. Και έτσι δεν ε, διακινδυνεύουμε τίποτα. Και το δεύτερο που θέλουμε να προβάλλουμε ως σοσιαλιστές είναι ότι δεν θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο ευθύ εξ αρχής να έχουμε αυτό το ε, στρώμα, το μαξιλαράκι ασφαλείας των 8 δις. Μπορεί να υπάρξει κάποια εξοικονόμηση σε κάποια γραμμή του προπολογισμού και να δούμε ότι να υπάρχει χρήμα εκεί. Αλλά θεωρούμε ότι 8 δις είναι υπερβολικό. Υπερβολική επιφυλακτικότητα. Είναι θέμα ρευστότητα. Γιατί ούτως ή άλλως ό,τι και να γίνει ο προπολογισμό εγγυείται 16 δις. Να βάλουμε ένα δις είτε έχουμε βάλει ένα δί ω αποθεματικό, είτε έχουμε βάλει πέντε, είτε έχουμε βάλει οχτώ δί ω αποθεματικό του ΕΦΣΥ. Ο προπολογισμό δίνει περισσότερε εγγύσεις από αυτό. Για παράδειγμα δίνει εγγύησει για τι εξωτερικέ δράσει ε, της Τράπεζας Επενδύσεων. Αλλά μπλοκάρουμε μόνο το 8 ή 9% εγγύσει στον προπολογισμό. Ο ευρωπαϊκό προπολογισμό εγγυάται και το μηχανισμό σταθερότητα. 60 δι. Και πόσο έχει μπλοκάρει ο προπολογισμό, 0. 0 γιατί η εγγύηση υπάρχει σε κάθε περίπτωση. Και αυτή είναι η βάση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Επενδύσεων. Εάν μειώσουμε το Ταμείο Εγγύσεων, διευκολύνουμε τον προπολογισμό, χρειαζόμαστε λιγότερα χρήματα να βρούμε σε πρώτη φάση και αν μετά τα χρειαστούμε, έχουμε την υποχρέωση να τα βρούμε. Δεν διακινδυνεύουμε λοιπόν τίποτα. Αυτά είναι τα δύο μηνύματα που θέλει να ε, τονίσει η σοσιαλιστική ομάδα. Ο κύριος Λούνης από το ECR. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα επαναλάβω τα όσα είπαν οι συνάδελφοι. Ούτω ή άλλω, κάποιε από τι παρατηρήσει μου είχα τη δυνατότητα να τι εκθέσω και σε προηγούμενε μα συνεδριάσει, να αναφερθώ σε τρία μόνο σημεία. Είναι σαφέ για όλου μα ποια είναι η θέση του ECR όσον αφορά τα βασικά ζητήματα. Καταρχά, θέλουμε κάποια προσωρινά κονδύλια, θέλουμε ως προς αυτό και έχουμε υποβάλει προς αυτό τροπολογίες στο κείμενο. Όπως είπαν και όλοι οι συνάδελφοι πριν από λίγο, θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Το ταμείο αυτό το ΕΦΣΥ δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για λόγους πολιτικούς. Δεν πρέπει να πολιτικοποιηθεί σε καμία περίπτωση. Αν εξετάσει όμω κανείς τις τροπολογίες των συναδέλφων, τελικά συνειδητοποιεί ότι όντως υπάρχουν κάποια θετικά στοιχεία στις τροπολογίες. Πρώτον, εμείς δεν θέλουμε πολιτικοποίηση όπως σας είπα. Αυτό σημαίνει ότι ε, ανησυχούμε πάρα πολύ για τους ελέγχους που μπορούν να γίνουν από τα κράτη-μέλη και ιδίως όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Επίσης, δεν θα θέλαμε να υπάρχει διοικητικό συμβούλιο. Παράλληλα όμως θα πρέπει να ενισχυθεί η Επιτροπή Επενδύσεων και να έχουμε ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες στην Επιτροπή αυτή. Και νομίζω ότι αυτό λένε και πάρα πολλές τροπολογίες και άλλων συναδέλφων. Για παράδειγμα, οι τροπολογίες 87, Εκεί πέρα μία συνάδελφος αναφέρεται ακριβώς σε μία επιτροπή επενδύσεων η οποία θα πρέπει να λειτουργεί εντελώς ανεξάρτητα. Στην 300 στην 838 με συγχωρείτε, βλέπουμε εδώ πέρα ότι θα πρέπει να γίνεται μια συγκεκριμένη ανεξάρτητη επιλογή επενδυτικών προγραμμάτων. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί συνάδελφοι οι οποίοι θέλουν αυτή την, προέφηση, την προσέγγιση. Και κάτι ακόμα. Θέλουμε να υπάρχει πραγματικά μια οικονομική προστιθέμενη αξία. Αν πραγματικά ιδιώτε επενδυτέ θέλουμε να συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό, προφανώ θα πρέπει να είναι ενδιαφέρον, θα πρέπει να είναι ελκυστικό για του ιδιώτε επενδυτέ. Και από την άλλη βλέπω ότι υπάρχουν ε, αρκετέ ε, τροπολογίε του κ. Χέκμαρ, για παράδειγμα, από το ΕΛΚ, που αναφέρεται και αυτό σε βιώσιμα επενδυτικά προγράμματα. Σε άλλε τροπολογίε αναφερόμαστε σε βιώσιμα προγράμματα από οικονομική πλευρά. Επίσης οι σοσιαλιστές αναφέρονται και αυτοί σε διατηρήσιμα βιώσιμα προγράμματα. Κύριε Γκουαλτιέρη, νομίζω ότι εσείς έχετε κάνει μια σχετική τέτοια τροπολογία. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε κεφαλιακή χρηματοδότηση χωρίς να υπάρχει πραγματικά μια βιώσιμη επένδυση από πίσω. Όπω είπε και ο κύριος Μπούλμαν, λοιπόν, πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβαστικέ λύσει, αλλά θα πρέπει να είναι σαφέ ότι για μα σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να δούμε πολιτικοποίηση αυτού του ταμείου. Καμία πολιτικοποίηση δεν πρέπει να λάβει χώρα και αυτό για μα είναι καθοριστικό. Και ολοκληρώνω Νομίζω ότι κάθε φορά που μιλάμε για το ΕΦΣΥ λέμε και θα πρέπει να λέμε ότι το Ταμείο αυτό δεν θα πρέπει να αποτελεί σε καμία περίπτωση εναλλακτική λύση όσον αφορά τι διαφορετικέ μεταρρυθμίσει και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να αποτελέσει μέσο δημοσίων επενδύσεων για τα κράτη-μέλη, δημόσια χρηματοδότηση για τα κράτη-μέλη. Σα ευχαριστούμε κύριε Λούνε. Όντω έχω υποβάλει τέτοιε τροπολογίε, οι οποίε λέω ότι όντω θα πρέπει να υπάρχει προσθετικότητα δεν ακριβώς αυτό το είπατε εσείς, αλλά χαίρομαι που σας άρεσε η τροπολογία μου. Ο κύριος Άσουαρτ είναι επόμενος ομιλητής, παρακαλώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω και εγώ κανένα δύο σχόλια. Πρόκειται για πρόγραμμα εφάνταστο και φιλόδοξο και πρέπει να σημειωθεί ότι χωρίς να πληρώνεται ούτε ένα ευρώ οι ανακοινώσεις της ΤΕΚ και της Κομισιόν ήδη έχουν αρχίσει να ε, δημιουργούν εμπιστοσύνη. Γι' αυτό θα στηρίξουμε ευρέως τη στάση του Συμβουλίου. Απ' την άλλη μεριά δεν πρέπει όλα αυτά να υπονομεύσουν το EMFF. Γιατί ορισμένοι συνάδελφοι θα πούν ότι είναι ευκαιρία να αυξηθούν τα κονδύλια του EMFF. Βέβαια όπως ξέρουμε καλά ο διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες και χρειάζεται περαιτέρω, χρειάζονται περαιτέρω διαβερτήσεις των λεπτομεριών. Επίσης ως παρατήρηση να προσέξουμε το εξής. Για την αναθέρμανση της ευρωπαϊκής οικονομίας χρειάζονται τρία πράγματα δηλαδή το, EF, και η ποσοτική χαλάρωση θα βοηθήσουν πολύ στη δημιουργία θέσεων απασχόληση, αλλά αυτό θα περιοριστεί, θα είναι περιορισμένο αν δεν εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνει το καθένα. Οι τροπολογίες που καταθέσαμε αποσαφηνίζουν ορισμένα στοιχεία της αρχικής πρότασης. Καταρχήν ξέρουμε ότι υπάρχει εδώ κάποιο ρίσκο και άρα τίθεται το θέμα των εγγυημένων χρηματοδοτήσεων όπως για αυτά που προβλέπει ο Ορίζον 2020. Έχουν κατατεθεί πολύ καλές τροπολογίες από συναδέλφους και τις έχω συστήσει και εγώ όποτε τις έχουμε συζητήσει. Απ' την άλλη τα δίκτυα διανομής πρέπει να γίνουν καλύτερα κατανοητά και τέλος όπως και άλλοι θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι για την κατανομή των ταμείων δεν πρέπει να γίνει πολιτικοποίηση. Θέλω όμως να τονίσω ότι θα ήταν σωστό και θεμητό το Κοινοβούλιο ως συνομοθέτης που άρα συνεκτίθεται στον κίνδυνο να έχει και αυτό κάποιο ρόλο για την επιτήρηση, την εποπτεία των αποτελεσμάτων. Ευχαριστώ. Ωραία. Από τους φιλελεύθερους ο κύριος Τρεμός. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα είμαι πολύ σύντομος, θα μιλήσω μόνο δύο λεπτά, γιατί άλλωστε έχουμε όλοι καταθέσει γραπτό στις τροπολογίες μας, να υπενθυμίσω τρεις βασικές ιδέες. Πρώτον, ξέρετε ότι οι φιλελεύθεροι και εγώ ως μεσογειακός φιλελεύθερος έχουμε μια κάποια αιμονία, θέλετε, σχετικά με μια σχετική προτεραιότητα. Νομίζω ότι ε, Πρέπει όλοι να συμφωνήσουμε ότι η προτεραιότητα λοιπόν θα πρέπει να δοθεί στα διασυνοριακά έργα. Κάθε φορά που θέλουμε να έχουμε ένα ευρωπαϊκό επενδυτικό σχέδιο, πρωταρχική θέση θα πρέπει να έχουν αυτά τα διασυνοριακά σχέδια και εφόσον θέλουμε να κινητοποιήσουμε ιδιωτικέ επενδύσει, θα πρέπει να προωθήσουμε την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία μέσω των προτινόμενων αυτών έργων. Δηλαδή, τα υποψήφια έργα θα πρέπει να δημιουργήσουν μια οικονομική και κοινωνική απόδοση, να δημιουργήσουν δηλαδή οικονομική ανάπτυξη και θέσει απασχόληση. Το έργο το οποίο κάναμε τελευταία πέντε χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε τώρα να το αξιοποιήσουμε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο τελευταία πέντε χρόνια αποφασίσανε πολύ συγκεκριμένα προγράμματα που έχουν να κάνουν με τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας. Νομίζω λοιπόν ότι ήδη τα τρία θεσμικά όργανα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Επιτροπή και Συμβούλιο, έχουμε ήδη την εμπειρία συζήτησης και έγκριση τέτοιων προγραμμάτων ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας στον τομέα, για παράδειγμα, των μεταφορών. Πρόκειται για διασυνοριακά έργα, τα οποία αξίζει να προωθήσουμε. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπενθυμίσουμε οι μεν στους δε ποια είναι τα έργα αυτά τα οποία εγκρίναμε στο παρελθόν. Νομίζω ότι τα έργα αυτά θα πρέπει να έχουν πρωταρχική θέση στα πλαίσια του Ταμείου αυτού. Διότι διαφορετικά πολύ φοβάμαι ότι σε πάρα πολλά κράτη-μέλη τα πράγματα θα συνεχίσουν όπως ακριβώς τώρα, χωρίς να γίνεται δηλαδή καμία θετική τροποποίηση, χωρίς να υπάρχει πραγματικά η βούληση για αυτή την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Business as usual δηλαδή. Μίλησα με συναδέλφου από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι οποίοι μου είπαν «Μα αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να εντοπίσουμε τίποτα, ούτε πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε συγκεκριμένα έργα». Αυτό ενδεχομένω να λειτουργήσει σωστά σε χώρε όπου ήδη γίνεται μια ανάλυση κόστου ωφέλους για την επιλογή τέτοιων προγραμμάτων. Αλλά καταλαβαίνετε ότι ελοχεύει πολύ σημαντικό κίνδυνο για τι χώρε εκείνε που δεν έχουν τέτοιο σύστημα. Ξέρετε ότι συζητήσαμε πρόσφατα και την έκθεση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και εκεί πέρα είδαμε ότι όντως υπήρχαν συγκεκριμένε ζημίες της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε σχέση με έργα για παράδειγμα της Ισπανίας τα οποία δεν είχαν υψηλό βαθμό διαφάνειας και που φάνηκε τελικά ότι χρησιμοποιήθηκαν κάποια κονδύλια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, τα οποία λαθασμένα χρησιμοποιήθηκαν, λαθασμένα επενδύθηκαν και οδήγησαν τελικά σε σημαντικές ζημίες για την ίδια την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αναφέρομαι σε έργα τα οποία ξεκίνησαν στην περιοχή της Καταλωνίας. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει πραγματικά να προωθήσουμε περισσότερο τα διασυνοριακά προγράμματα και τα προγράμματα ευρωπαϊκής προστιθέμενης αξίας. Ξέρω ότι ε, με αιμονή έχω αναφερθεί πολλά και στο παρελθόν στο ζήτημα αυτό, αλλά δυστυχώς καμία άλλη πολιτική ομάδα δεν το έχει αναφέρει. Πολύ θετική λοιπόν η εργασία των ε, συνεισηγητών. Νομίζω λοιπόν ότι μέσω και των τροπολογιών μπορούμε να βελτιώσουμε περισσότερο το κείμενο και να ανταποκριθούμε τελικά στους πολίτες εκείνους που ζητούν περισσότερη Ευρώπη, περισσότερη και καλύτερη Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ ο συμπρόεδρος. Σε ευχαριστώ Ρομπέρτο. Ο κύριος Τόρβαλς λείπει νομίζω, επομένως το λόγο έχει η κυρία Νηριάντα. Λίγα λόγια από την ΚΟΕ. Θέλω να ευχαριστήσω τους συζητητές που έκαναν πολύ καλή δουλειά και φυσικά θα χρειαστεί και πολύ περισσότεροι. Όπως και οι άλλοι ομιλητές δεν θα επαναλάβω τα πάντα. Εμένα με ενδιαφέρει ιδιαίτερα το θέμα της επίπτωσης στον προϋπολογισμό και θα υποστηρίξω τις τροπολογίες που αφορούν αυτό το θέμα ιδιαίτερα για τους συνεταιρισμούς και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ιδίως οι κοινωνικές επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί δεν θέλουμε να μπουν σε δεύτερη μοίρα και αυτό νομίζω ότι πρέπει να γνωρίζουμε ανα πάσα στιγμή ότι οι επενδύσεις πρέπει να κατευθυνθούν στις, στους τομείς όπου χρειάζονται περισσότερο. Για την έρευνα και την καινοτομία ξέρουμε, βλέπουμε ότι πρέπει να είναι κινητήρια δύναμη της αναδέρμανσης και ξέρουμε ότι σε αυτό υπάρχουν ελλείψεις στον ορίζοντα 2020 και για την ε, κατανομή των κοντιλίων από το ΕΦΣΥ. Πρέπει βέβαια να υπάρχει και λογοδοσία και διαφάνεια και όλες οι τροπολογίες που ζητούν αυτόν τον στόχο θα στηριχθούν από μας καθώς και η προσβασιμότητα και βέβαια ποιοτικός έλεγχος οι περιφέρειες που δεν θα συμπεριληφθούν στις επενδύσεις ίσως θα έπρεπε να συμπεριληφθούν σύμφωνα με ορισμένα κριτήρια <clears throat> οι τροπολογίες λοιπόν που στηρίζουν και διασφαλίζουν την ε, κάλυψη αυτών των ελλημάτων θα στηριχθούν και αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Λείπει ο κύριος Δεμάζη νομίζω. Ο κύριος Βάλλη λοιπόν. Ο κύριος Δεμάζη απουσιάζει, έτσι δεν είναι, ο κύριος Φάμπιο Δεμάζη. Το λόγο έχει ο κύριος Μαραγκά, λοιπόν. Ah, Ούτως ή άλλως εκπροσωπούμε και τις διεπιτροπές, ε, και την ΕΚΟΝ και την ε, Budget. Λοιπόν, αντικαθιστάτε λοιπόν τον κύριο Έικουτ. Έχετε λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα αγγλικά. Δεν θα επαναλάβω το ότι συμφωνούμε προφανώς ότι θα πρέπει να τονώσουμε περισσότερο τις επενδύσεις στην Ευρώπη και απευθυνόμενος και στον κύριο Λούνες πρέπει να πω ότι οι επενδύσεις μπορούν να οδηγήσουν σε διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Ενδεχομένως να μην συμμεριζόμαστε τις δικέ σας όσον αφορά το είδος των διαφορετικών μεταρρυθμίσεων, αλλά χρειαζόμαστε προφανώς επενδύσεις προκειμένου να τονώσουμε τις διαφορετικές μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη. Τα δύο λοιπόν συνδέονται άμεσα. Έχουμε κάποιες αμφιβολίες όμως όσον αφορά τη μέθοδο που θα ακολουθηθεί από το επενδυτικό αυτό σχέδιο. Πολλές φορές η προσέγγισή μας είναι αρκετά αισιόδοξη, ιδίως όσον αφορά το επίπεδο της χρηματοδότησης και πολλές φορές νομίζουμε ότι το ίδιο το πρόγραμμα είναι αρκετά μικρό όσον αφορά τις επενδύσεις που θέλουμε να πετύχουμε. Όσον αφορά τώρα τις τροπολογίες μας, νομίζω ότι πρέπει να στοχεύουμε κυρίως σε επενδύσεις, όχι όμως με πολιτικό τρόπο, αλλά λαμβάνοντα υπόψη την πραγματική προστιθέμενη αξία για την οικονομία. Ως προς αυτό λοιπόν εμείς θα θέλαμε να κατευθύνουμε περισσότερο τις επενδύσεις προς την Στρατηγική Ευρώπη 2020 και τους στόχους που έχουμε εκεί, ακριβώς επειδή μπορεί να έχουμε οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές θετικές συνέπειες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να συνάδει περισσότερο το σχέδιο το επενδυτικό αυτό με τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Θα πρέπει επίσης να κατευθύνουμε επίση τις επενδύσεις εκεί όπου μπορούμε πραγματικά να αντιμετωπίσουμε περισσότερο μέσω επενδύσεων το χάσμα παραγωγικότητας που έχει εντοπιστεί. Δεν νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε άδικα επενδύσεις σε τομείς που δεν χρειάζεται να γίνουν επενδύσεις, αλλά να επικεντρωθούμε περισσότερο στο χάσμα παραγωγικότητας, τροπολογία 740. Αναφερόμαστε επίση και στι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Μέχρι στιγμή βλέπουμε ότι οι μεγάλε επιχειρήσει έχουν πρόσβαση στι κεφαλαγορές, έχουν πρόσβαση σε επενδύσεις. Δεν είναι αυτές που πρέπει να βοηθηθούν, Κυρίω οι μικρομεσαίες επιχειρήσει πρέπει να στηριχθούν και συμφωνώ με του προλύσαντε ότι και κοινωνικέ επιχειρήσει θα πρέπει να υποφεληθούν από το επενδυτικό αυτό σχέδιο. Επίση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων δεν θα πρέπει να επενδύσει τεχνολογίε του παρελθόντο για παράδειγμα σε παλαιές μορφές ενέργειας όπως ο άνθρακας, τα ορυκτά καύσιμα κτλ. Νομίζω θα πρέπει να κρατηθούμε περισσότερο στις ε, νέες τεχνολογίες, οι μορφές ενέργειας του μέλλοντος. Και συμφωνώ με τον κύριο Άσχουαρθ ότι δεν θα πρέπει οι ε, νομοθέτες, οι πολιτικοί να διαχειριστούν το πρόγραμμα αυτό. Από την άλλη εμείς δεν θέλουμε να δώσουμε και λευκή επιταγή. Θεωρούμε λοιπόν ότι στα πλαίσια του ε, κανονισμού ΕΦΣΥ θα πρέπει να διευθετούνται τα περισσότερα πράγματα με τον κανονισμό, αλλά θα πρέπει στη συνέχεια να έχουμε και καταξιοδότηση πράξης, προκειμένου να μπορούμε κάποιες λεπτομέρειες να τις αποφασίζουμε εκτός κανονισμού. Αλλά για όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχει και κατάλληλη εποπτεία και ο κατάλληλος έλεγχος. Επίση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει πρόσβαση σε ενημέρωση και πληροφορίε και θα πρέπει να υποβάλει επίση ερωτήματα όσον αφορά την στρατηγική αυτή κατεύθυνση του επενδυτικού προγράμματο. Και ω προ αυτό δεν θέλουμε λευκή, επιταγή και αυτό το λόγο υποβάλαμε σχετική τροπολογία. Επίση, θέλουμε τακτικέ αναφορέ για του υπεύθυνου του ΕΦΣΥ προκειμένου να υπάρχει μια διασύνδεση ανάμεσα στην ανάληψη δράση και τι επιπτώσει που έχει δράση αυτή να βλέπουμε δηλαδή ποιο είναι ο πραγματικό αντίκτυπο από τι επενδύσει του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Και κατά αυτόν τον τρόπο θα δούμε κατά πόσο πραγματικά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το σχέδιο αυτό, κατά πόσο είναι ρεαλιστικό. Επίση θα πρέπει να διασφαλίσουμε την σωστή λειτουργία του Ταμείου και πώς θα λειτουργούν επίσης οι τυχόν διαμεσολαβητές. Επίσης, θα πρέπει να μπορεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχει περισσότερο στο διορισμό του διευθύνοντας, του Διευθύνοντα Συμβούλου και να πληρωτεί Διευθύνοντα Συμβούλου όσον αφορά την Επιτροπή Επενδύσεων. Όσον αφορά τώρα την προέλευση τη χρηματοδότηση, αυτό που μα προκαλεί μια κάποια ανησυχία είναι ότι όσον αφορά τον κοινοτικό τουλάχιστον προπολογισμό, αυτή τη στιγμή παίρνουμε χρήματα από τα τμήματα κίνητου προπολογισμού που ήδη κατευθύνονται προ τι επενδύσει. Δηλαδή, η διευκόλυνση συνδέοντα την Ευρώπη και ορίζοντα 2020 είναι από μόνο του επενδυτικά προγράμματα. Θα ήταν πιο λογικό να παίρναμε χρήματα από άλλα τμήματα του κοινοτικού προπολογισμού ή ακόμα και από το φυστάμενο περιθώριο ευελιξία που υπάρχει στα πλαίσια του προπολογισμού. Ανταυτού βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι παίρνουμε χρήματα από επενδυτικά προγράμματα του κοινοτικού προπολογισμού, τα οποία ήδη φύστανται και ήδη έχουν θετικά αποτελέσματα. Επίσης, ε, θεωρούμε ότι η συμφωνία θα πρέπει να υπογράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να χρησιμοποιούνται κατεξοδοτήσει πράξεις, αλλά να μπορούμε να έχουμε και εμείς ως νομοθέτες έλεγχο επ' αυτού Βλέπουμε πολλές φορές πως λειτουργούν ε, διάφορες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως η Κίνα. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα πρέπει να αποφύγουμε όμως τέτοια μοντέλα. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε έναν κεντρικοποιημένο χαρακτήρα διαχείρισης του προγράμματος αυτού. Αντίθετα, θα πρέπει να υπάρχει και μια κάποια αποκέντρωση. Είναι σημαντικό να μπορούμε να έχουμε δηλαδή και συμμετέχονται σε τοπικό, περιφερειακό επίπεδο προκειμένου τα επενδυτικά αυτά προγράμματα πραγματικά να έχουν έναν οικονομικό αντίκτυπο, να οδηγήσουν σε οικονομική προστιθέμενη αξία. Όσον αφορά τώρα την Επιτροπή Επενδύσεων, τον έχουμε μόνο οικονομολόγου ή ανθρώπου από το χρηματοπιστωτικό τομέα σε αυτή την Επιτροπή Επενδύσεων δεν είναι θετικό. Αυτή τη στιγμή θέλουμε να δημιουργήσουμε προστιθέμενη αξία για τι κοινωνίε. Οικονομική, κοινωνική, περιβαλλοντική προστιθέμενη αξία. Γι' αυτό το λόγο θα θέλαμε η Επιτροπή Επενδύσεων να αντικατοπτρίσει τη σύνθεσή τη και του στόχου αυτού. Και τέλο, και αυτό αποτελεί μεγάλη ανησυχία για τη δική μου πολιτική ομάδα, με την υφιστάμενη διάρθρωσή του, φοβόμαστε τελικά ότι το Ταμείο αυτό ενδεχομένω να μην καταφέρει να ωφελήσει τι χώρε και τι περιφέρειες εκείνες που το χρειάζονται περισσότερο. Ιδίω όσον αφορά τους κανόνες συγχρηματοδότησης. Μας προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης όπως ισχύουν σήμερα θα αποτρέψουν ορισμένα κράτη-μέλη από το να έχουν πρόσβαση στο σχέδιο αυτό προκειμένου να καταφέρουν και τέτοια να συγχρηματοδοτήσουν επενδυτικά προγράμματα. Θα θέλαμε λοιπόν περισσότερη ευελιξία στο Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη, προκειμένου να κατευθύνουμε τελικά τι επενδύσει εκεί που πραγματικά τι χρειαζόμαστε. Ευχαριστώ πολύ. Merci, monsieur Ευχαριστώ κύριο Μαραγάλ. Να συνεχίσω τη γραμμή σκέψης του Φιλίπ Λαμπέρ. Το ΕΦΣΙ έχει ένα πρόβλημα αξιοπιστίας υπόθηκε και από τους εισηγητές. Πρέπει λοιπόν να τους δώσουμε, να του δώσουμε τη μέγιστη αξιοπιστία. Γι' αυτό κύριο στόχος των τροπολογιών μας είναι να περιγράψουμε τα προγράμματα που θα θέλαμε να χρηματοδοτηθούν από το ΕΦΣΥ. Είναι σημαντικό να συμβάλλει σε μια πιο βιώσιμη Ευρώπη. Θέλουμε λοιπόν σαφή κριτήρια. Για παράδειγμα, η καταπολέμηση των αερίων θερμοκηπίου, ανανεώσιμες, εκπαίδευση, κατάρτιση, αλλά και προγράμματα σε περιφέρειες με χαμηλό εισόδημα, υψηλή ανεργία. Όχι λοιπόν προγράμματα που δεν πληρούν αυτούς τους στόχους. Επειδή είναι λίγοι πόροι, πρέπει να υπάρχει σαφής προσθετικότητα. Πρέπει επίσης η Τράπεζα Επενδύσεων να λάβει υπόψη και τα θέματα ισότητας φύλων. Η Αφρικανική Τράπεζα Επενδύσεων και η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων έχουν σαφείς πολιτικές για αυτό το θέμα. Και πρέπει και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να έχει τέτοια προγράμματα τέτοια κριτήρια, συγγνώμη. Αλλά από πού λοιπόν θα έρθουν οι χρηματοδοτήσεις. Συμφωνούμε με εκείνους που λένε ότι στο μέτρο του δυνατού πρέπει να διατηρηθούν οι χρηματοδοτησει συμφωνουμε με εκεινου που λενε οτι στο μετρο του δυνατου πρεπει να διατηρηθουν οι χρηματοδοτησει του συνδεοντα στην Ευρώπη και του ορίζον 2020 να αξιοποιήσουμε τα υπάρχοντα περιθώρια και την ευελιξία στον υπάρχοντα προπολογισμό, όπω είπε η κυρία Γαρδιά Θάβαλ προηγουμένω. Και γιατί όχι. Τα ετήσια πλεονάσματα του προπολογισμού. Πολύ σημαντικό μέσω χρηματοδότηση. Βεβαίω, να συζητήσουμε τη δυνατότητα διαφορετική χρήση πόρων. Για παράδειγμα, πόρου από το ΙΤΕΡ. Αλλά και άλλα, και άλλες περιπτώσεις όπου μπορεί να γίνει επανα, νέα χρήση. Για παράδειγμα και στην κοινή γεωρική πολιτική, μέσω ανώτατου ορίου της ε, πληρωμής προς τις εκμεταλλεύσεις ή κάποιες ε, υποχρεώσεις από την προηγούμενη περίοδο των προοπτικών της πολιτικής ε, συνοχής. Βέβαια είναι πολύ περίπλοκο το θέμα και πολύ δυσχερές λόγω της ε, δημοσιονομικής συγκυρίας. Αλλά μπορούμε να αξιοποιήσουμε και το αποθεματικό για τα απρόβλεπτα αν μείνουν χρήματα. Λοιπόν, καλύτερα να λαμβάνονται σε ετήσια βάση αποφάσεις. Και αυτό έχει υποθεί. Επίσης, πρέπει να δίδεται αποκεντρωμένη βοήθεια. Και όχι μόνο βοήθεια, αλλά πραγματική συμμετοχή των ε, εμπλεκομένων φορέων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Διότι υπάρχουν εταιρικέ σχέσεις στα πλαίσια της λειτουργίας των διαθροτικών ταμείων. Θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για τα προγράμματα του ΕΦΣΙ συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το ρόλο που μπορεί να έχει για το, την Επιτροπή Εποπτείας και τον ε, επικεφαλής του Ταμείου. Και εδώ πρέπει να το δούμε. Βεβαίως η Επιτροπή Επενδύσεων πρέπει να έχει τους κατάλληλους εμπειρογνώμονες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι μόνο χρηματοδοτικές, χρηματοπιστωτικές οι πλευρές αποτίμησης των προγραμμάτων. Χρειαζόμαστε λοιπόν ιδιωτικές επενδύσεις. Αν τι θέλουμε δεν πρέπει να θέτουμε πολλές προποθέσει. Αλλά πρέπει να υπάρχει ισχυρή, ισχυρός έλεγχος. Το Κοινοβούλιο πρέπει να πει ότι πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό ούτω ώστε οι ιδιωτικοί επενδυτές να έχουν ίδιο συμφέρον για να βοηθήσουν για να δημιουργηθεί ανάπτυξη, απασχόληση και να μειωθούν οι περιφερειακές ανισότητες που είναι η πραγματική αιτία τόσο πολλών κρίσεων που έχουμε αντιμετωπίσει στο κοινωνικό και οικονομικό τομέα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Λείπει ο κύριος Βάλλη νομίζω. Ζάνη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο ε, και να θίξω μόνο τα σημεία εκείνα τα οποία θεωρώ ότι είναι σημαντικά για μα, για τη δική μα πολιτική ομάδα. Άλλωστε, οι συνάδελφοι έχουν αναλύσει εκτενώ όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Πρώτο, λοιπόν, ε, όσον αφορά τη διακυβέρνηση. Εγώ δεν είμαι τόσο πεπισμένο ε, ότι θα πρέπει να αποκλείσουμε την πολιτική διάσταση από το Ταμείο αυτό. Το Ταμείο αυτό αποτελεί πολιτική απόφαση, πολιτική επιλογή. Επομένω, θα πρέπει να υπάρχει απαραίτητη πολιτική εγγύηση ότι όντω μέσω του Ταμείου αυτού προσπαθούμε να ακολουθήσουμε και να πετύχουμε κάποιου στόχου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων δεν νομίζω ότι έχει ακολουθήσει του στόχου αυτού στο παρελθόν και όντω είδαμε ότι υπήρχαν ε, και κάποια προγράμματα τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων όπω το πρόγραμμα Κάστορ στην ε, Ισπανία ή ε, άλλα προγράμματα στην Ιταλία τα οποία εσφαλμένα χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τελικά οδήγησαν σε ζημίες. Ακριβώς λοιπόν για αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια πολιτική διάσταση και θα πρέπει στο Τεχνικό Συμβούλιο να υπάρχει ένας εκπρόσωπος από κάθε κράτος μέλος, ο οποίος θα εγγυάται ότι όντως το Ταμείο αυτό ακολουθεί και εξυπηρετεί τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και για πρόθεση της πράσινης ενέργειας και οικονομίας όσον αφορά τη δημοκρατική λογοδοσία. Και αυτό το ζήτημα είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει τόσο με τη διακυβέρνηση όσο και με τι επενδύσει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ω μοναδικό θεσμικό όργανο το οποίο εκλέγεται άμεσα από του πολίτε, θα πρέπει προφανώ να μπορεί να έχει ένα δημοκρατικό έλεγχο για αυτό το ταμείο. Θα πρέπει να δίνει τον τελικό λόγο έγκριση όσον αφορά τον διορισμό τη Επιτροπή Επενδύσεων, η οποία θα κληθεί να αξιολογήσει και να εγκρίνει όλα τα προτινόμενα υποψήφια προγράμματα. Όσον αφορά τώρα την τυπολογία των επενδύσεων, νομίζω ότι θα πρέπει εν μέρη να ασχοληθούμε με το τμήμα εκείνο του ταμείου το οποίο θα χρηματοδοτεί υποδομές και ένα άλλο τμήμα του Ταμείου που θα χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι υπάρχει ένας ισότιμος διαχωρισμός ανάμεσα στα δύο. Εμείς θα θέλαμε το Ταμείο αυτό να προωθεί περισσότερο τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν πραγματικά τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας. Σε αυτές θα πρέπει να καταφέρουμε να εστιαστούμε. Επίσης τις νεοσύστατες επιχειρήσεις, τις startup εκείνες οι οποίες πραγματικά συμβάλλουν πάρα πολύ στην δημιουργία της απαραίτητης υποδομής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και προωθούν επίσης και την καινοτομία και κατ' επέκταση όχι μόνο την οικονομία αλλά και την ίδια την κοινωνική ανάπτυξη. Όσον αφορά τα κριτήρια τα επενδυτικά, το ανέφεραν αυτό και οι συνάδελφοι. Νομίζω ότι ως προς αυτά θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να προωθήσουμε τους τομείς εκείνους ή τις περιοχές εκείνες μάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη καθυστέρηση επενδύσεων εξαιτία οικονομικής κρίσης. Αν θέλουμε να έχουμε μια ενιαία Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ενιαία ταχύτητα αν θέλετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να εστιάσουμε τις επενδύσεις αυτού του Ταμείου στις περιοχές Ευρωπαϊκής Ένωσης που υστερούν περισσότερο. Ως προς αυτό λοιπόν εμείς θα θέλαμε να υπάρχει μια μεγαλύτερη εμπλοκή και από τους τοπικούς περιφερειακούς παράγοντες, από την τοπική πολλές φορές αυτοδιοίκηση, η οποία γνωρίζει πολύ περισσότερο πού βρίσκονται τα επενδυτικά κοινά, ποιες είναι οι περιφέρειες που στερούν περισσότερο, προς τα πού θα πρέπει να διοχετευτούν οι επενδύσεις. Ένα ακόμα σημείο, το ζήτημα της διαφάνειας. Ζήτημα πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως ε, υπό το φως των κριτηρίων διαφάνειας που δημοσίευσε πρόσφατα τις τελευταίες εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Ανησυχώ κάπως γιατί... Ε, λίγες εβδομάδες προτού τεθεί ε, ισχύει το Ταμείο αυτό, τα κριτήρια διαφάνειας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων πραγματικά δεν είναι επαρκή, είναι εντελώς επιφανειακά. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει πραγματικά να υπάρχουν αυστηρά κριτήρια διαφάνειας όσον αφορά την επιλογή επενδύσεων στα πλαίσια αυτού του Ταμείου. Όσον αφορά τώρα την εγγύηση, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούμε να συμφιλιώσουμε τον στόχο διασφάλισης μιας βιώσιμης υποστήριξης για να καταφέρουμε να προσελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσεις, μέσω δηλαδή μιας εγγύησης και πώς από την άλλη θα καταφέρουμε σε αιτήσια βάση να χρηματοδοτούμε το Ταμείο Εγγύησεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι εξ αρχής θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ένα σημαντικό ποσό για την εγγύηση, θα πρέπει να γνωρίσουμε από πού θα χρηματοδοτεί η εγγύηση αυτή, από πού θα προέρχονται οι πόροι, προκειμένου αυτό να χρησιμοποιηθεί ως σημαντικό κίνητρο για να προσελκύσουμε επενδύσεις. Αν δεν γίνει κάτι τέτοιο, πολύ φοβάμαι ότι θα δημιουργηθεί μία αβεβαιότητα για τους ιδιώτες επενδυτές, οι οποίοι θα θεωρούν ότι θα υπάρχει απαραίτητη ευρωπαϊκή εγγύηση και δημιουργείται και μία αβεβαιότητα όσον αφορά και τον ίδιο τον προπολογισμό. Ξέρετε ότι ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάθε φορά να καταφέρουμε να δούμε από πού θα προέλθουν οι πόροι. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θεωρώ ότι εξ αρχής από την αρχή του ταμείου αυτού θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη βεβαιότητα όσον αφορά τη χρηματοδότηση της εγγύησης. Γι' αυτό κατ' επέκταση θα οδηγήσει σε πιο σίγουρες επενδύσεις στο μέλλον. Θα καθησυχάσει δηλαδή αυτό τους επενδυτές. Εύχομαι ότι θα έχουμε μια πολύ θετική συνεργασία με τις υπόλοιπε πολιτικές ομάδες. Εύχομαι καλό κουράγιο σε όλους. Πιέζει ο χρόνος και η δουλειά που μας περιμένει είναι πολύ δύσκολη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ακούσαμε τους δύο εισηγητές λοιπόν και τους σκιώδεις. Τώρα θα αρχίσει η συζήτηση. Ποιοι θέλουν το λόγο. Κυρία Τωμά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συζητητές και να τους εκφράσω όλοι μας την ηθική και πολιτική στήριξη. Καταρχήν συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος Καράς και η κυρία Γκουαρντία Σαμπάλ ως προς τη θέληση του Κοινοβουλίου να καταλήξει με τις προτινόμενες διορίες και προθεσμίες αλλά και με την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα που θέλουμε να εγγυηθούμε. Υπάρχουν ακόμη μερικά εκκρεμή σημεία για μένα, τρία θα αναφέρω, για να βελτιωθεί η λειτουργία του Ταμείου αυτού. Πρώτον, ως μέλος της Επιτροπής Προϋπολογισμών θα ήθελα να μιλήσω για τις επιπτώσεις που θα έχει επί του προϋπολογισμού των δημοσιονομικών μας. Ότι συνδέεται το Ταμείο αυτό με τον προϋπολογισμό είναι καταρχήν και καθεαυτό μια σημαντική εγγύηση. Δεν έχουμε πρόβλημα λοιπόν με αυτή τη σύνδεση, αλλά για τη θέση του προϋπολογισμού που επελέχθηκε αυτή μας φαίνεται προβλεπτική και το έχουμε πει πολύ. Παραδείγματος χάρη, οι προβλέψεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας δείχνουν ότι υπάρχουν προβλήματα, θα υπάρξουν προβλήματα με τον ορίζοντα 2020 ως προς την έρευνα. Η δημοσιονομική ευελιξία νομίζω ότι επιτρέπει βέλτιστη στάθμιση και Πιστεύω ότι είναι λάθος να λέμε ότι μπορεί να προσθεθεί εδώ αστάθ, αβεβαιότητα για τους επενδυτές διότι το Ταμείο Εγγύσεων συνδέεται με τον προϋπολογισμό ακριβώς άρα η σταθερότητα είναι απόλυτη το μόνο θέμα είναι ποια επιλογή θα γίνει όπως είπε και η κυρία Γορδία Ζαβάλ ποιες δυνατότητες μας επιτρέπει ο προϋπολογισμός αλλά κίνδυνος δεν υπάρχει και επίσης συμφωνώ να μην πειράξουμε τα 16 δισεκατομμύρια του Ταμείου Εγγύσεων αντίθετα την επιλογή του 50% της σύνδεσης του προϋπολογισμού με τον προϋπολογισμό νομίζω ότι αυτή είναι αυθαίρετη το ίδιο αυθαίρετη με το 3% του ελλείμματος που είχε προβλεφθεί για τους δημόσιους προϋπολογισμούς θα μπορούσαμε να πούμε ότι συνδέεται όχι κατά 50, κατά 30, κατά 25, δεν αλλάζει όμως αυτό τίποτα ως προς τον μηχανισμό. Αυτό ήταν το πρώτο. Δεύτερον τώρα, τι όρους βάζουμε. Είπαμε να μην μπλοκαριστούν ή αποκλειστούν ορισμένες κατηγορίες προγραμμάτων γιατί δεν θέλουμε να ξεχάσουμε τους αρχικούς και κυρίους στόχους μας όπως την απασχόληση γιατί γι' αυτό, σχεδόν μόνο γι' αυτό δημιουργείται αυτό το επενδυτικό ταμείο και άρα να μην τεθεί αυτό σε κίνδυνο. Εξάλλου θυμίζω ότι η σύνδεση με τον ορίζοντα 2020 ή το Connecting Europe μπορεί τελικά να μην αποδειχτεί προσθετική. Και συμφωνώ με αυτό που λέει και το άρθρο 5 για την προστιθέμενη αξία ως προς το περιβάλλον και τα κοινωνικά. Τώρα η θέση των περιφερειών και των τοπικών τραπεζών. Επ' αυτού κατέθεσα τροπολογίες. Γιατί όχι μόνο για την αποκέντρωση αλλά και γιατί έχει αποδειχτεί ότι οι περιφέρειες και οι τοπικές επενδυτικές τράπεζες είναι αυτές που επιτόπου συνδέονται με τη ζωή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τα προγράμματα, τα σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι εκείνα που δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις εργασίας και άρα με τις τροπολογίες αυτές επιζητώ μια βελτίωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεπρέ ο οποίος ε, είναι ο του κ. Νίλ που είναι σκιώδη συγητής, αλλά Επιτροπή Επιτροπής Προπολογισμού, αλλά θα εκφραστεί προσωπικά ο κ. Ντεπρέ. Ευχαριστώ. Ναι, αντικαθιστώ τον κύριο Τόρβαντ που είναι σκιώδης ε, της ομάδας Άλτε. Με συγχωρείτε που καθυστέρησα. Είχα κάποια προβλήματα σήμερα το πρωί. Λοιπόν, να τονίσω πρώτα το εξή. Το εύση που προτείνει ο κύριος Γιούνκερ είναι ένα νέο μέσο. Ένα νέο μέσο δεν πρέπει να περιέχει όλα τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά των προγραμμάτων που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Αυτό που είναι καινούριο πρέπει να αντιμετωπιστεί καινοτόμα όχι πάντα σε όλα τα νέα εγχειρήματα στοιχεία που ε, περιλαμβάνονται σε άλλα εγχειρήματα που χρηματοδοτώνται αλλιώς. Πρώτο αυτό. Για τα κριτήρια λοιπόν ως συμπέρασμα. Τα κριτήρια για την επιλογή των προγραμμάτων θα πρέπει πρώτον να επιφέρουν προσθετικότητα. Αυτό δεν είναι θέμα σύγκλησης. Θα πρέπει λοιπόν αυτό το νέο ταμείο να χρηματοδοτήσει προγράμματα που δεν θα χρηματοδοτούνταν με τα παραδοσιακά μέσα. Και δεύτερον να είναι υψηλού κινδύνου. Και τα εγχειρήματα υψηλού κινδύνου κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι πτώση θα έχουν στην απασχόληση. Για παράδειγμα, όταν έγιναν οι πρώτε έρευνε που οδήγησαν ε, στο ίντερνετ, αν τους ρωτούσαμε πόσες ε, θέσεις εργασίας θα δημιουργούνται, δεν θα ξέραν να απαντήσουν. Και ξέρουμε τα αποτελέσματα. Συμβάλλει τόσο πολύ και στην ανάπτυξη και στην απασχόληση το ίντερνετ. Να αποφύγουμε λοιπόν κριτήρια που δεν μπορούν να συνδυαστούν με τους στόχους του Ταμείου. Βεβαίω. οι στόχοι του Ταμείου πρέπει να συνδυάζονται με του γενικού στόχους της Ένωσης. Σε αυτό συμφωνούμε. Τρίτον, αν θέλουμε όντως να δώσουμε κάθε δυνατότητα σε αυτό το Ταμείο να επιτύχει ως καινούριο πρόγραμμα, οι μηχανισμοί του θα πρέπει να είναι εντελώς ανεξάρτητοι από πολιτικές παρεμβάσει. Κάποιοι συνάδελφοι άκουσαν να συμμετέχουν ε, στη Διοικητική Επιτροπή εκπρόσωποι των κρατών μελών. Τι θα γίνει δηλαδή, θα πρέπει να υπάρχει δίκαια επιστροφή, να έχουν όλο εκεί πέρα σαν τσοπανόσκυλα να λένε «Α, στη χώρα μου δεν έχουν δοθεί επαρκείς χρηματοδοτήσεις, άρα δεν ε, εγκρίνω». Γιατί οι περιφέρειες που εκπροσωπώ δεν έχουν λάβει αρκετές χρηματοδοτήσεις. Μα αυτό είναι αντελώ αντίθετο από τη λογική του νέου αυτού ταμείου για να παίξει κάποιο ρόλο. Γι' αυτό λοιπόν, για τον ίδιο λόγο της μη πολιτικής παρέμβασης, είμαστε επιφυλακτικοί παρά το ότι το προτείνουν δύο συγητές, τον οποίο χαιρετίζω εμπαρόδο την εργασία. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε επιφυλάξεις με το ρόλο που θα παίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τον καθορισμό κάποιων των και εμπειρογνωμόνων. Δεν είναι δυνατόν μια κοινοβουλική επιτροπή να κρίνει την ποιότητα των ε, εμπειρογνωμόνων που θα αποφασίσουν για προγράμματα με τι κριτήρια. Το παρελθόν τους, ε, την πολιτική τους τοποθέτηση, αυτά που θα μας πούνε. Μα με τι κριτήρια θα αποφασίσουμε κάτι τέτοιο. Πώς θα έχουμε τέτοια δυνατότητα. Δεν βλέπω πραγματικά, δεν καταλαβαίνω πώς θα το κάνουμε. Και δεν νομίζω ότι είναι δική μας δουλειά αυτό. Δική μας δουλειά είναι να λειτουργεί με συνέπεια αυτό το μέσο, να έχει την αναγκαία χρηματοδότηση Λοιπόν, θέλω να είμαι ιδιαίτερα επιφλακτικός και για τις τροπολογίες που προτείνουν οι δύο εισηγητές όσον αφορά τις παρεμβάσεις του Κοινοβουλίου στην επιλογή των εθνόντων και σε κάθε περίπτωση στην επιλογή των εμπειρογνωμόνων. Αυτό θεωρούμε ότι είναι απόλυτα ανεφενίας για την πρικοδότηση τώρα. Κοιτάξτε, το ουσιώδες για όλους τους ενδεχόμενους επενδυτές δεν είναι με τι τρόπο θα χρηματοδοτήσουμε το ταμείο. Είναι ότι θέλουν μια εγγύηση ότι αυτό το ταμείο εγγυήσεων θα έχει επαρκή χρηματοδότηση για να δίνει εγγυήσει. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Πέρα από όσα θα δώσει η Τράπεζα Επενδύσεων, συνολικά η εγγύηση αυτή να είναι στο ύψος 16 δις και τα 8 δις να περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό. Ξέρω ότι ορισμένοι έχουν επιφυλάξει από αυτού, εμείς δεν έχουμε. Θεωρούμε ότι 8 δί είναι το κατάλληλο ποσό. Τώρα, πώς λοιπόν θα προοικοδοτηθεί αυτό το ταμείο. Συμφωνώ με όλους όσους είπαν και νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση ότι δεν είναι δυνατόν να συμφωνήσουμε με την πρόταση της Κομισιόν. Να πάρουμε δηλαδή από τον ορίζοντα 2020 και το μέσο συνδέοντα την Ευρώπη. Αυτό που πρέπει να είναι η κατεύθυνσή μας είναι ότι κάθε χρόνο θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε για να είναι επαρκώς χρηματοδοτημένο το Ταμείο, αλλά θα το κάνουμε πριν θίξουμε τα δύο προαναφερθέντα προγράμματα, εξαντλώντας τις άλλες δυνατότητες που μας προσφέρει ο προπολογισμό και υπάρχουν αρκετές. Και σε ορισμένους, επειδή ξέρω ότι ανησυχούν ορισμένοι, θέλω να τους πω το εξή. Γιατί ορισμένοι λοιπόν έλεγα θεωρούν ότι αν δεν λάβουμε υπόψη, αν δεν ε, συμπεριλάβουμε τα άρθρα 18-19, μειώνουμε την αξιοπιστία των εγγύσεων καθόλου. Δεν είναι τα άρθρα 18 και 19 που θα μας κάνουν να αποφύγουμε την, ε, τον ετήσιο χαρακτήρα του προπολογισμού. Κάθε χρόνο, ανεξάρτητα από το μηχανισμό χρηματοδότησης, η Κομισιόν ή εμείς να έχουμε την πρωτοβουλία να βάλουμε στον προπολογισμό τις αναγκαίες χρηματοδοτήσεις. Το 18 και 19 μας εκείνονται μόνο ότι θα τα πάρουμε από τον ορίζοντα 20, 2020 και το συνδέοντα στην Ευρώπη. Και αυτό δεν το θέλουμε, αλλά κατά τα άλλα, εφόσον τονίσουμε ότι θα δώσουμε σε αυτό το εύση όσα χρειάζεται, ούτω ή άλλω οι μηχανισμοί ετησιότητα του προπολογισμού επιβάλλουν του ίδιου περιορισμού. Δεν πρέπει λοιπόν να υποκύψουμε στου εκβιασμού κάποιων στην Επιτροπή ή αλλού που λένε δεν θα έχει καμία αξιοπιστία το Ταμείο εάν δεν συμπεριλάβεται τα άρθρα 18 και 19. Τελευταίο, Πρόεδρε, για το οποίο δεν έχουμε καταλήξει πλήρως σε άποψη. Διερωτώμεθα, η συμφωνία μεταξύ της Τράπεζας Επενδύσεων και της Επιτροπής θα πρέπει να έχει τη μορφή κατεξοδότηση πράξης. Υπάρχουν υπέρ και κατά. Υπέρ, αν θυμάμαι καλά, διότι είναι μια τεχνική που γνωρίζουμε. Αλλά υπάρχουν και κατά. Δηλαδή, στις κάτι εξοδότηση πράξη υπάρχει κάποια αβεβαιότητα ότι κάποια στιγμή το Κοινοβούλιο έχει τη δυνατότητα να λήξει την ισχύ μιας κατεξοδότηση πράξης, να την ακυρώσει. Και τι κατάσταση θα δημιουργήσει αυτό. Πριν λοιπόν ε, επιλέξουμε αυτή τη λύση, να το συζητήσουμε μεταξύ μας σε βάθος για να δούμε αν και κατά πόσο είναι σκόπιμο. Γιατί υπάρχει τρόπος να εγγυηθούμε και τη διαφάνεια και το κοινοβουλευτικό έλεγχο με τον καλύτερο τρόπο χωρίς κατανάγκη να περάσουμε από αυτή τη λύση. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρος. Ο κύριος Σδροζεύσκη. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, εγώ είμαι εισηγητής για την Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού Πρόκειται για την ε, επιτροπή αυτή, η οποία αντιστοιχεί τελικά σε ένα πολύ μικρό ποσό των ε, προβλεπόμενων επενδύσεων. Πάντως έχει καθοριστική σημασία το της παιδείας και του πολιτισμού να αφορά την ίδια την επιτυχία του επενδυτικού σχεδίου. Ξέρετε ότι ε, αυτή τη στιγμή ασχολούμεθα με διάφορα έργα, με διάφορα προγράμματα, τα οποία Θέλουμε να δούμε πώς θα καταφέρουν να τύχουν υλοποίηση στα πλαίσια του Ταμείου αυτού. Πολλές φορές βλέπουμε ότι ορισμένοι θέλουν απλώς μέσω του Ταμείου αυτού να υποστηρίξουν τα όσα έχουν επιτευχθεί στα πλαίσια του κοινοτικού προπολογισμού. Ανταυτού νομίζω ότι θα πρέπει οι στόχοι μας να ήταν πολύ πιο συγκεκριμένοι. Προκειμένου να επιτύχει οικονομικά η Ευρώπη, θα πρέπει να έχει υψηλή ανταγωνιστικότητα, ένα απλό φορολογικό σύστημα, ενεργειακή ασφάλεια όσον αφορά τον εμβοδιασμό και μια κοινή ενεργειακή πολιτική εν τέλει. Καθώς συζητούμε λοιπόν για το ταμείο αυτό, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, και μάλιστα στα πλαίσια της όλης συζήτησης που γίνεται για τους ελάχιστους μισθούς, τα ελάχιστα, τις αποδοχές για τους οδηγούς φορτηγών, θα έλεγα ότι υπάρχουν πραγματικά πάρα πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί κανείς να τονώσει τις επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μόνος πάντως τρόπος ε, για να επιτύχουμε και οικονομικά είναι να μην δημιουργήσουμε περαιτέρω επιπλοκές στη λειτουργία της ενίας αγοράς. Και αυτό θα έλεγα ακριβώ ω βασικό επιχείρημα και βασικό μέλημα για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Χαιρετίζω λοιπόν το καταπληκτικό έργο που έχουν κάνει οι δύο εισηγητές. Θα έλεγα όμως ότι θα έπρεπε τουλάχιστον να υποβληθούν κάποιε ε, ελάχιστε τροπολογίε, μικρό αριθμό τροπολογιών, προκειμένου να μην περιπλέξουμε περισσότερο την έγκριση αυτού του ταμείου. Κυρία Μούντι, έχει το λόγο. Κλέρ Μούντι, παρακαλώ. Uh, yes. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου του συζητητέ για την εργασία που έχουν κάνει και για την εργασία που καλούνται να κάνουν βέβαια στο μέλλον. Θα ήθελα όμω να πω κιόλα και ακούγοντα του προαλήσαντε, ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να καταφέρει να καταλήξει γρήγορα σε μια συμφωνία και βλέπουμε βέβαια ότι καθυστερούμε. Βλέπουμε από την άλλη όμως ότι έχουν υποβληθεί τροπολογίες οι οποίες παρουσιάζουν μια κάποια σύγκληση και που τελικά οδηγούν στην βελτίωση του κειμένου προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να καταλήξουμε σε ένα μηχανισμό ο οποίος είναι πραγματικά αποτελεσματικός. Θα οδηγήσει δηλαδή σε αυτό που θέλουμε όλοι, οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δύο συγκεκριμένα πράγματα τώρα. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όντως θα υπάρχει προσθεθικότητα Δηλαδή δεν θα πρέπει να πάρουμε κονδύλια από τομείς που ήδη δημιουργούν οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρομαι προφανώς κυρίως στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 και βέβαια δεύτερον θα πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος ότι όντως επιτυγχάνουμε τους ευκταίους στόχους μέσω αυτού του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει εξ αρχής να έχουμε ξεκάθαρα κριτήρια και θα πρέπει στη συνέχεια να έχουμε την απαραίτητη ενημέρωση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη δυνατότητα βέβαια να κάνουμε αξιολόγηση του αντικτύπου. Να δούμε δηλαδή αν όντως πιάνουν τόπο οι επενδύσεις αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Μόσκα έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να προσθέσω κι εγώ μόνο κάποιες σύντομες παρατηρήσεις γιατί νομίζω τα περισσότερα πράγματα έχουν ήδη υποθεί από τους συναδέλφους. Να ξεκινήσω από ένα ζήτημα το οποίο με αφορά ιδιαίτερα. Όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, έτσι και εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε μέσω του Ταμείου αυτού να τονώσουμε την οικονομική ανάκαμψη ως κράτη, ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ακόμα και ως θεσμικά όργανα. Ιδίω κατά τη διάρκεια μιας περίοδου που βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα αξιοπιστία για τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω λοιπόν το Ταμείο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί κυρίως προκειμένου να καταφέρουμε να ενισχύσουμε την προσπάθεια αυτή. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην βελτίωση της προβολής του Ταμείου αυτού και εξάντε και εξπόστα. Προβολή δηλαδή του Ταμείου αυτού προκειμένου να γίνει κατανοητό ότι το εγχείρημα αυτό, το Ταμείο αυτό μπορεί τελικά να έχει άμεσες θετικές επιπτώσεις στη ζωή όλων των πολιτών και σε όλε τι επιχειρήσει Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή νομίζω ότι πρέπει να είναι, αν θέλετε, η βασική φιλοσοφία η οποία, βάσει τη οποία θα πρέπει στη συνέχεια να δούμε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να πάρει το ταμείο αυτό και ποιε επενδύσει θα μπορούσαμε να προωθήσουμε και ποιε θα πρέπει να είναι τροποποιήσει που θα γίνουν στη λειτουργία του ταμείου. Θα πρέπει το βασικό μα μέλημα να είναι να ανακτηθεί η εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων πολιτών. Τώρα να περάσω σε κάποιε λεπτομέρειε. Συμφωνώ και εγώ ότι θα πρέπει να έχουμε πάντα κατά νου το κριτήριο της προσθετικότητας, σε σχέση δηλαδή με τις επενδύσεις που θα πρέπει να υλοποιηθούν, αλλά θα πρέπει να πετύχουμε πάντα την κατάλληλη εξισορρόπηση ανάμεσα το ότι θα πρέπει να κάνουμε μεν επενδύσεις, αλλά θα πρέπει οι επενδύσεις αυτές, τα έργα αυτά να είναι και βιώσιμα στη συνέχεια, να είναι διατηρήσιμα. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει και αυτή η απαραίτητη κοινοτική εγγύηση προκειμένου το Ταμείο αυτό να μπορεί να λειτουργήσει βιώσιμα, σε βάθος χρόνου δηλαδή. Δεύτερη παρατήρηση. Με ενδιαφέρει ιδιαίτερα η αναφορά που έγινε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στις ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί προσταθήσαμε να κάνουμε και μία επιπλέον αναφορά όχι μόνο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και στις λεγόμενες μικροεπιχειρήσεις αλλά επίσης και στα δίκτυα μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Γιατί ξέρετε ότι πολλές φορές τα δίκτυα αυτά ή ο τρόπος που εμφανίζονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που λειτουργούν διαφέρει από τη μία χώρα στην άλλη. Πιστεύω λοιπόν θα πρέπει να καταφέρουμε μέσω του ταμείου αυτού να εμπλέξουμε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μπορούν δηλαδή όλες να υποφεληθούν. Επίσης, είναι σημαντικό να δώσουμε έναν πιο βελτιωμένο ορισμό όσον αφορά τις ε, διασυνοριακές λειτουργίες, ε, συναλλαγές, επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτό άλλωστε αφορά πάρα πολλέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η διασυνοριακή συνεργασία. Θα πρέπει να καταλάβουμε περισσότερο λοιπόν τι εννοούμε όταν λέμε διασυνοριακέ επιχειρήσει, cross-border operations, προκειμένου να καταφέρουμε τελικά να βοηθήσουμε και τις χώρες εκείνες οι οποίες ε, χρειάζονται περισσότερες επενδύσεις. Κατά αυτόν τον τρόπο νομίζω ότι θα γίνουν πιο συνεκτικές και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα αφορούν όλες τις χώρες της Ένωσης. Νομίζω θα πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι διαφορές που υφίστανται ανάμεσα στις χώρες της Ένωσης. Και χωρίς να γίνουμε πάρα πολύ αυστηροί όσον αφορά τα κριτήρια της, του περιφερειακού χαρακτήρα των επενδύσεων, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν χώρε στι οποίε υπάρχει σημαντική επενδυτική καθυστέρηση, σημαντικό επενδυτικό κενό και θα πρέπει και οι χώρε αυτέ να καταφέρουν να έχουν καλύτερη πρόσβαση. Πρόκειται για χώρε οι οποίε πλήττονται από οικονομική καθυστέρηση, από υψηλότατα ποσοστά ανεργία. Θα πρέπει λοιπόν κάπου στο κείμενο να γίνεται μία αναφορά και στι χώρε αυτέ. Και μια τελευταία παρατήρηση νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και το είπανε και αυτό και οι συνάδελφοι, να έχουμε καλύτερη διασύνδεση του Ταμείου αυτού με τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις. Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, ιδίως θα θέλουμε να βελτιώσουμε κάποιους από τους ορισμούς που χρησιμοποιούνται στο προτινόμενο κείμενο. Ευχαριστώ, δεν βλέπω να θέλει κανείς άλλο το λόγο. Οπότε να ζητήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που εκπροσωπείται από τον κύριο Μπενχαμίν Άνχελ να μας ενημερώσει για την άποψή της ε, μετά από όλα όσα υπόθηκαν. Ευχαριστώ και τον κύριο Άνχελ και τη μαγκερία Μαρία Σόμπαραγκάν που εκπροσωπεί την ΕΤΕ και που θα πάρει το λόγο μετά τον κύριο Άνχελ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω κυρίως πέντε θέματα προϋπολογισμό, διακυβέρνηση, κρατικές επιχορηγήσεις, αναφορές και άλλα. Αρχίζω με τον προϋπολογισμό όπου βλέπω ότι υπάρχουν ακόμη διαφορές απόψεων στο Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν είναι απολύτως πεπισμένη ότι το Κοινοβούλιο δεν πρέπει απλώς να καταργήσει το χρηματοδοτικό σχέδιο λέγοντας ότι θα αφαιθεί στην ετήσια συζήτηση επί του προϋπολογισμού. Όχι. Μια τέτοια απόφαση μπορεί να είναι και παράνομη αυτή τη στιγμή εφόσον το άρθρο 310 της συνθήκης ρητά μας υποχρεώνει να διασφαλίσουμε ότι κάθε διευθέτηση που θα εγκριθεί θα συμφωνεί με το ΠολΔΙΠ και αυτό δεν προβλέπει τα 8 δισεκατομμύρια. Ας μην επαναλάβω το επιχείρημα που άκουσα στο Στρασβούργο την περασμένη φορά για τα, τις επιπτώσεις που θα έχουν όλα αυτά στη δυνατότητά μας προβλεψιμότητας των ευρωπαϊκών δαπανών θα ήθελα απλώς να αναφέρω άλλα στοιχεία. Μερικοί αναρωτήθηκαν γιατί δεν παίρνουμε τα λεφτά προσθέτοντας το 1 δις, το 1 αυτό θα σήμαινε αλλαγή του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και όπως ξέρετε αυτό είναι πολύ λεπτό και επικίνδυνο θέμα. Το να πάρουμε χρήματα από το αποθεματικό των διαρθρωτικών ταμείων δεν θα άλλαζε μόνο το πολδίπ, αλλά θα, δεν θα άλλαζε μεν το πολδίπ, αλλά θα άλλαζε άλλες διατάξεις του επενδυτικού ταμείου και σας υπενθυμίζω ότι ο, κανονισ... ο σχετικός κανονισμός έγινε μετά από 67 τριμερείς διαλόγους. 67. Επομένως το να ανοίξουμε αυτό το κουτί θα σήμαινε ότι ανοίγουμε κουτί της Πανδώρας. Το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο είναι σαφές ότι το εργαλείο ευελιξίας από την άλλη, όπου ανέφεραν πολλοί από εσά, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί παρά μόνο μέσα σε έναν ενιάυσιο χαρακτήρα εξέτασης του προπολογισμού αφού έχουν εξαντληθεί όλες οι άλλες δυνατότητες και άρα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολυετή χρηματοδότηση όπως συζητάμε τώρα. Άρα μόνο το ένα α μπορούμε να προσθέσουμε και αυτό σημαίνει ότι η κατάσταση είναι πολύ σαφής. Αν θέλουμε τον ορίζοντα 2020 και το Connecting Europe να τα στηρίξουμε περαιτέρω, να τα αυξήσουμε, τότε θα εργαστούμε να περικόψουμε άλλα προγράμματα, όπως τον έρασμο. Θέλει το Κοινοβούλιο να γίνουν τρομερές περικοπές στον έρασμο. Τώρα για το μέγεθος του Ταμείου Εγγύσεων Α, όχι, όχι, δεν ε, κάνω κανέναν εκβιασμό. Σας αναφέρω τα προγράμματα που συμπεριλαμβάνει το 1α. Έρασμος Γαλιλαίο Φισκάλη. Μικρά, μικρού ύψου είναι όλα αυτά, αλλά το Horizon 2020 και το Connecting Europe είναι το 70% του 1α. Λοιπόν, για το Ταμείο Εγγυήσεων Τρία πράγματα χρειάζονται. Πρώτον, να διασφαλιστεί προσθετικότητα. Το είπαν και αυτό πολλοί από εσά. Είναι κοινό στόχος της Κομισιόν του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Και για να διασφαλιστεί η προσθετικότητα πρέπει να υπάρξουν πλαίσια που να μας επιτρέπουν ανάληψη περισσότερου κινδύνου. Αν αρχίσουμε μειώνοντας το ύψος του ταμείου αυτού τότε δεν ξέρουμε πια τι εννοεί να κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά, τι σημαίνει. Δεύτερον, πρέπει να υπάρχει προβλεψιμότητα στον προϋπολογισμό. Όπως γνωρίζετε, η στάθμιση του κινδύνου που έγινε από την ΕΤΕ και την Κομισιόν κατέληξε ότι υπάρχει κίνδυνος απώλειας 6,5 δισεκατομμυρίων. Μερικοί από εσά μπορεί να λένε γιατί να μην μειώσουμε το ταμείο στα 6,5 δισεκατομμύρια λοιπόν. Θα σας έλεγα ειλικρινά ότι αυτό είναι μια πρόβλεψη με βάση στατιστικές πιθανότητες απλώς και ότι μόνο στην πράξη μπορούμε να δούμε τι απώλειες μπορεί να έχουμε πραγματικά. Είμαστε δε πεπισμένοι για αυτόν τον λόγο ότι πρέπει να υπάρξει κάποιο είδους ενδιάμεσο ποσό για να μην έχουμε εκπλήξεις και καταλήξουμε ξαφνικά σε κανένα δημοσιονομικό δράμα. Τελευταίος λόγος, η περικοπή ή μάλλον όχι. Ακούστηκαν ήδη πολλά για το ότι πολύ λίγα δημόσια χρήματα μπήκαν σε αυτό το σχέδιο. Εγώ δεν είμαι βέβαιος πώς θα ερμήνευε ο τύπος την απόφαση να μειωθεί το συνολικό ποσό. Μερικοί από εσά επίσης όπως και ο κύριος Φερνάντες πρότειναν ότι ξεπερνάει το Ταμείο Εγγυήσεων να διατεθεί αλλού. Αυτό μπορούμε να το εξετάσουμε, αλλά έχει επίσης τονιστεί ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρξει κάποια λεγόμενη ρήτρα του ραντεβού. Και αυτό μπορούμε να το επανεξετάσουμε με το, μαζί με το Κοινοβούλιο. Για τη διακυβέρνηση παρακαλώ να προσέξετε τον πειρασμό οι κατευθυντήρες γραμμές των επενδύσεων να βασιστούν κυρίως σε κατεξουσιοδότηση πράξης. Όλοι γνωρίζουμε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο υπάρχει ο κίνδυνος να έχουμε αντιρρήσεις και σχόλια και από όλες τις χώρες μέλη και τις βουλές. Και τελικά θα καταλήξουμε σε ένα πολύ μια πολύ υπερφορτωμένη διαδικασία και ατέλειωτες συζητήσεις. Τώρα καταλαβαίνω βέβαια ότι μερικά από αυτά που είπατε εννοούν να μην δοθεί λευκή επιταγή στην ΕΤΕ και στην Κομισιόν. Πρέπει λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να διασφαλιστεί ότι θα έχετε τις πληροφορίες που χρειάζεστε. Για τη δυνατότητα συμμετοχής στο ΕΦΣΥ και στο Διοικητικό του Συμβούλιο με τους εκπροσώπους ιδιωτικού τομέα και των κρατών η Κομισιόν δεν αποκλεί αυτή την πιθανότητα, απλώς δεν είναι και τίποτε πρωτόγνωρο. Υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις όπου ο ιδιωτικός τομέας συμμετέχει μαζί με τον δημόσιο σε τε, ανάλογα ταμεία, όπως στο μελλοντικό επενδυτικό. Παρ' όλα αυτά, αν το Κοινοβούλιο θέλει, πρεσβεύει όπως και το Συμβούλιο, ότι καλύτερο είναι να περιοριστεί η συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο φυσικά τότε η Κομισιόν μπορεί να το δεχτεί και να το λάβει υπόψη της για την Επενδυτική Επιτροπή και την προηγούμενη φορά σας είχα πει ότι έχουμε ανησυχίες για την πολιτικοποίηση της, ε, του ορισμού των μελών αυτής της Επιτροπής. Πρέπει να είναι όλα τα μέλη πλήρως ανεξάρτητα. Αυτό είναι ο ακρογωνίος λήθος των προτάσεών μας. Αν αμφισβητηθεί η ανεξαρτησία οποιοδήποτε, μπορεί τελικά να μην πετύχουμε τίποτα και να μην επιτευχθεί κυρίως το 80% ιδιωτικών επενδύσεων που ζητάμε. Πρέπει να προσέξουμε λοιπόν ιδιωτικής χρηματοδότησης μάλλον. Όπως είπε και ο κύριος Ντεπρέ, εμπειρογνώμονας μόνο μπορεί να ορίσει άλλον εμπειρογνώμονα. Εγώ ασχολούμαι με το επενδυτικό σχέδιο από το Σεπτέμβριο και δεν είμαι σε θέση, δεν θα ήμουν σε θέση να επιλέξω τον κατάλληλο εμπειρογνώμονα. Πρέπει να ρωτήσουμε, να ζητήσουμε την άποψη ανθρώπων που είναι και οι ίδιοι εμπειρογνώμονες. Άλλοι είπαν να ενισχυθεί η ανεξαρτησία αυτής της Επιτροπής. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση και θα μπορούσαμε να συνεργαστούμε ώστε ο κανονισμός να ενισχυθεί ως προς την ανεξαρτησία της Επιτροπής αυτής. Εκφράσατε την ανησυχία ότι αν υπάρχει το σωστό μείγμα δικαιοδοσιών και εμείς το συζητούμε αυτό πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει απαραίτητη γνώση των διάφορων γεωγραφικών και άλλων διαφορών της αγοράς και θέλουμε να συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο ώστε η σύνταξη του κανονισμού να είναι τέτοια ώστε να το διασφαλίζει. Για τον ε, διοικητή εμείς δεχόμαστε αυτό που είπατε για τις δικαιοδοσίες του και καταλαβαίνουμε ότι ανάλογα με ό,τι αποφασίστηκε πέρυσι για διάφορα καινούργια προγράμματα είμαστε διατεθειμένοι να συνεργαστούμε και γι' αυτό. Για τις περιφέρειες και τις τοπικές επενδυτικές τράπεζες που ανέφεραν πολλοί από εσά. πράγματι δεν υπάρχει συγκεντρωτισμός το σχέδιο. Οποιοςδήποτε επενδυτής μπορεί να υποβάλει σχέδιο αν κριθεί ότι το σχέδιο αυτό είναι βιώσιμο και δεν μπορεί να εφαρμοστεί με άλλο τρόπο χωρίς την ενωσιακή εγγύηση θα σταλεί στην Επενδυτική Επιτροπή η οποία θα γνωμοδοτήσει καταλήλως αλλά δεν υπάρχει απριόρι περιορισμός στα σχέδια ως προς το τι θα εξεταστεί από την ΕΤΕ ας πούμε. Οποιοςδήποτε ιδιώτης μπορεί να υποβάλει το σχέδιό του και θα εξεταστεί αρμοδίως. Για τις κρατικές επιχορηγήσεις ή βοήθειες ξέρουμε ότι και αυτό είναι σημαντικό θέμα. Εμείς στην Κομισιόν ακόμη προετοιμάζουμε τις κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές επιχορηγήσεις ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι ό,τι γίνει θα συμβαδίζει με τα ισχύοντα για τις κρατικές επιχορηγήσεις. Και δεν θα επιβάλλουμε, δεν θα επιβαρύνουμε ιδιαίτερα τα πράγματα για να μην καθυστερήσει η εφαρμογή του σχεδίου. Αλλά απ' την άλλη θέλουμε συνοχή και συνέπεια σε ό,τι προβλεφθεί με προηγούμενες αποφάσεις. Ας πούμε να μην υπάρχει επικάλυψη για τις υποδομές ή υπερβολική αντιστάθμιση πέρα από αυτήν που θέλουμε ούτως ή άλλως να πετύχουμε. Λόγω δε της δοκιμής αυτής που θα κάνουμε για τη συνέπεια και συνοχή ως προς τις κρατικές επιχορηγήσεις θα μπορέσει να γίνει επιτάχυνση τελικά της εφαρμογής. Σήμερα αν ένα κράτος θέλει να συγχρηματοδοτήσει ένα σχέδιο χρειάζεται περίπου ένας χρόνος για να εγκριθεί αυτή η συγχρηματοδότηση. Η Επενδυτική Επιτροπή όμως με τις ε, εξετάσεις που θα κάνει θα μπορεί μόνο σε δύο μήνες, σε δύο μήνες μόλις να δίνει το πράσινο φως για τέτοιες επιχορηγήσεις. Άρα θα επιταχυνθεί η διαδικασία σε σχέση με την τωρινή. Τώρα για την αξιολόγηση και τις αναφορές που απαιτούνται, λάβαμε υπόψη μας όσα μας είπατε για αυτά, καθώς και για την πληροφόρηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλες αυτές τις τροπολογίες που μιλούν για αυτά θα τις εξετάσουμε με θετικό πνεύμα. Για τη διάρκεια του Ταμείου, όπως ξέρετε η Κομισιόν, παρακαλώ να τελειώνετε κυρία μου, Α, τέλειωσε εγώ λοιπόν. Η Κομισιόν λέει το Ταμείο να είναι αϊθαλές. Στις συζητήσεις μας με το Συμβούλιο φάνηκε ότι τα κράτη-μέλη κινούνται μάλλον προς την κατεύθυνση που είπατε και εσείς δηλαδή ότι πρόκειται για κάτι καινούργιο και γι' αυτό χρειάζεται πολύ πλήρης αναθεώρηση μετά από, αξιολόγηση μετά από τρία χρόνια για να δούμε αν χρειαστεί τότε να αλλάξει τίποτα. Θέμα κοινή λογικής μου φαίνεται. Και καταλήγω ευχαριστώντας τα μέλη του Κοινοβουλίου για το τεράστιο ενδιαφέρον που επέδειξαν για το σχέδιο αυτό σχεδόν 2.000 τροπολογίες αυτό δείχνει ότι είναι προτεραιότητα και για μας και για σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και λυπούμε αν μακρηγόρησα τυχόν. Ευχαριστώ κύριε Άγχελ. Βεβαίως όσα είπατε μας ενδιαφέρουν. Ε, να καθησυχάσω τους συζητητές θα πάρουν τον λόγο. Ο κύριος Μπέγκε όμως είχε μια αντίδραση. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ένα... Έχω μεγάλη εκτίμηση για την ε, σοφροσύνη της Κομισιόν. Αλλά η αλαζονία με την οποία παρουσιάζει τις θέσει δεν με βρίσκει καθόλου σύμφωνο. Φυσικά υπάρχουν το άρθρο 310. Το άρθρο 310 υπάρχει και το, ο ετήσιος χαρακτήρας του προπολογισμού και το θέμα του πώς θα αξιοποιήσουμε τα 2,1 που δεν έχουν αξιοποιηθεί είναι θέμα, γιατί είναι στα πλαίσια της ε, ετήσιας διαδικασίας του προπολογισμού έχουμε τον κανόνα ότι θα έχουμε ένα ε, βαθμό ευελιξίας συν, 10, πλην 10%. Δηλαδή όλα αυτά θέλετε να τα καταργήσετε. Γιατί θεωρείτε ότι δεν ε, εγγυόμαστε αρκετά τα 8 δις. Θέλουμε να τα εγγυηθούμε, αλλά θέλουμε να είναι σαφή διαδικασία. Οπότε να συμβουλευτούμε. Κοιτάξτε τι έχουμε διαπραγματευτεί στο παρελθόν. Κοιτάξτε τι έχουμε κάνει στο παρελθόν με τη συμφωνία και της Κομισιόν του Γαλιλαίων, για το ΊΤΕΡ, για το μέσο, για τα τρόφιμα ή για το πακέτο συγκυρίας. Εάν συνεχίσετε να δράτε όπως κάνετε, τότε χάνουμε χρόνο και εσείς θα φταίτε που δεν θα τηρήσουμε τις ε, προθεσμίες. Να μιλείτε με τον τρόπο σας και να μην ξαναπείτε τέτοια πράγματα. Ευχαριστώ κύριε Μπέγκε. Η κυρία Μαρία Σομπέργεν της Τράπεζας Επενδύσεων. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους Ευρωβουλευτές για τη δυνατότητα που μας δίνετε να παρευρεθούμε σήμερα, να ακούσουμε τις απόψεις σας και για τη στήριξη που δίνετε στην Τράπεζα Επενδύσεων για να είναι ο διάβλος για την ε, διοχέτευση των πόρων του ΕΦΣΥ. Και την παίρνουμε πολύ σοβαρά αυτή την ευθύνη. Θέλουμε να το ξέρετε. Όταν σας άκουγα, μου ήρθε στο νου μια φράση που λένε τα παιδιά μου. Να μειώνουμε, να ξαναχρησιμοποιούμε και να ανακυκλώνουμε. Να μειώσουμε λοιπόν ε, την πρόσβαση σε δημόσιους πόρους. Παράλληλα προωθώντας επενδύσεις. Περί αυτού πρόκειται. Θέλουμε, αύξηση και θέλουμε ανάπτυξη και απασχόληση και θέλουμε μακροχρόνια ανταγωνιστικότητα για την Ένωση να μειώσουμε τη χρήση πόρων ε, ενώ προωθούμε τις επενδύσεις. Να ξαναχρησιμοποιήσουμε, τι εννοώ, αυτό το κεφάλαιο σποράς που με βάση την ανάλυση σας ελπίζω θα συμφωνήσετε να χορηγήσετε τα 16 δις στην ΕΤΕ για το Ταμείο Εγγύσεων εμείς θα συμβάλλουμε 5 δις από το δικό μας κεφαλιακό δυναμικό και έτσι θα έχουμε δυνατότητες να χρηματοδοτήσουμε πολλά. Η ΕΤΕ θα συμβάλλει 60 δις ρευστού από εμά, χάρη σε εγγυήσει και χάρη στο τριπλό Α που έχουμε ω πιστοληπτική ικανότητα, θα, θα μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε τα κεφάλαια στι αγορέ. Και η άλλη συμβολή τη ΕΤΕ θα είναι η δυνατότητα να εφαρμόσει τα προγράμματα. Όλο μα το προσωπικό θα αφιερωθεί σε αυτή την προσπάθεια. Και τι θα ανακυκλώσουμε τώρα. αλλάζουμε τον τρόπο αντιμετώπισης. Αντί να δίνουμε επιχορηγήσεις, δίνουμε δάνεια. Και αντί για επιδοτήσει, δίνουμε εγγυήσει. Όλα αυτά είναι επιστρέψιμα. Να θίξω τρία θέματα. Και εκτιμώ πολύ τις απόψεις για τρία θέματα κλειδιά. Το πρώτο είναι ότι η εγγύηση που δίνεται στην ΕΤΕ πρέπει να είναι ρωμαλαία Χαίρομαι πολύ για αυτό που είπατε, χωρίς προϋποθέσεις και αμετάκλητη. Είναι ζωτικό αυτό. Επίσης, οι πληρωμέ μέσω του Ταμείου Εγγύσεων πρέπει να γίνονται στην ώρα τους. Εγκαίρως. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη ότι αυτή η εγγύηση δεν θα πρέπει να κατακαιρματιστεί. Πρέπει να δοθεί στην ΕΤΕ αυτή η εγγύηση και η ΕΤΕ θα εργαστεί με του εθνικού οργανισμού και τις τράπεζες ε, για την προώθηση των επενδύσεων και με τις κλαδικές πλατφόρμες. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ποιος είναι σε τελευταία ανάλυση αρμόδιος για να προκύψουν τα 315 δις. Και γι' αυτό αρμόδιοι είναι η ΕΤΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να μην κατακαιρματίσουμε λοιπόν ε, τη λογοδοσία. Να λάβουμε υπόψη ότι στόχος μας είναι να προωθήσουμε τις ενωσιακές πολιτικές και όχι κατά περίπτωση εθνικά συμφέροντα, να μην ε, συμβάλλουμε κι εμείς στον κατακαιρματισμό των χρηματαγορών. Αυτό οπωσδήποτε δεν θα βοηθήσει την αξιοπιστία του εγχειρήματός μας. Τώρα για την προσθετικότητα. Και αυτό πολύ σημαντικό στοιχείο. Έχουμε συνέστηση ότι για μας, για την ΕΤΕ δεν είναι η συνηθισμένη δουλειά μας. Αυτό το ξέρουμε ξέρω ότι θέλουμε να χρηματοδοτήσουμε προγράμματα που δεν θα χρηματοδοτούνταν με του συνηθισμένου όρου. Όχι εκεί που δεν είναι καθόλου δυνατή χρηματοδότηση. Γιατί δεν υπάρχει καμία χρηματοδότηση, καμία δυνατότητα χρηματοδότηση. ίσω αυτό να σημαίνει πω δεν πρέπει να υπάρξει. Αλλά θέλουμε να προωθήσουμε προγράμματα που δεν χρηματοδοτούνται με τι συνήθει διαδικασίε και κριτήρια. Επειδή κρατάει πάρα πολύ χρηματοδότηση, Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλέ μικρομεσαίε επιχειρήσει οι οποίε πρέπει να περιμένουν ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναφέρομαι λοιπόν σε μικρομεσαίε επιχειρήσει οι οποίε μπορεί να έχουν τη μορφή startups και θα πρέπει να καταφέρουμε να τι συνοδεύσουμε σε όλη την εξέλιξή του. Α μην ξεχνάμε ότι οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι ο βασικό εργοδότη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ότι ε, στα 4 ευρώ τα οποία θα κινητοποιήσουμε τουλάχιστον ένα θα πάει στι μικρομεσαίε επιχειρήσεις και αυτό θα γίνει μέσω του Ευρωπαϊκού Αυτού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Επίσης, ποιο είναι το δίκτυο κατανομής, ήταν μια ερώτηση. Μα κοιτάξτε, είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Το δίκτυο αυτό θα πρέπει να ενδυναμωθεί, αλλά θα γίνει μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Πάντως το δίκτυο αυτό διανομής ήδη υπάρχει και είναι αξιόπιστο. Όσον αφορά την προσθετικότητα, Πρέπει να σας πω ότι προφανώς χρειαζόμαστε έργα τα οποία θα πρέπει να επιλεγούν βάσει της οικονομικής τους αξίας, της δυνατότητας να οδηγήσουν σε οικονομική απόδοση και τη δυνατότητά τους να έχουν κοινωνικές και περιβαλλοντικές θετικές επιπτώσεις. Ως Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων γνωρίζουμε πολύ καλά το ζήτημα αυτό. Χρηματοδοτούμε περίπου 500 έργα ετησίως. Θα πρέπει μέσω του νέου αυτού ταμείου να χρηματοδοτήσουμε επιπλέον 100-150 έργα. Έχουμε όμως ήδη την εμπειρογνωμοσύνη. Ας ε, χρησιμοποιήσουμε λοιπόν την εμπειρία μας αυτή, τη γνώση μας αυτή, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Όσον αφορά τώρα τη διακυβέρνηση, για μας το σημαντικό είναι η διακυβέρνηση αυτή να είναι απλή, λιτή και να μην δημιουργεί επιπλέον επίπεδα πολυπλοκότητος, αν θέλετε, όσον αφορά την διοίκηση. Όσον αφορά το Steering Board, το Διοικητικό Συμβούλιο, θεωρούμε ότι είναι εξορρεπημένη η πρόταση. Για την Επιτροπή Επενδύσεων συμφωνούμε με εσά ότι θα πρέπει η επιλογή των εμπειρογνωμών να γίνει σε μια τεχνική βάση και ότι χρειάζεται βέβαια και ευρύ εκπροσώπηση πολλών διαφορετικών τομέων αλλά και εθνικοτήτων. Πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε μια συμβολή σε διάφορους τομείς γνώσης που υπάρχει αυτή τη στιγμή η Επιτροπή Επενδύσεων θα πρέπει να έχει μία εντολή που ουσιαστικά θα συνδέεται με τη χρησιμοποίηση του Ταμείου Εγγύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται να κάνει την επιλογή των προγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι αυτή που θα επιλέγει τα προγράμματα και θα χρηματοδοτεί τα προγράμματα αυτά με την υποστήριξη της κοινοτική εγγύησης. Θα λογοδοτεί βασικά για την επιλογή των προγραμμάτων η ίδια η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να ολοκληρώσω λέγοντα τα ακόλουθα. Πρώτον, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή επιγόντω να δοθεί νέα τόνωση για τι επενδύσει. Δεν μπορούμε να χάνουμε χρόνο και εκτιμούμε βέβαια όλε τι προσπάθειε που έχουν καταβάλει οι Ευρωβουλευτέ και οι υπηρεσίε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ανάλογε προσπάθειε καταβάλει και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προφανώ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι προγράμματα τα οποία δεν χρηματοδοτούνταν στο παρελθόν θα αρχίσουν πλέον τώρα να χρηματοδοτούνται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Δεύτερη και τελευταία παρατήρηση. Θα πρέπει προφανώς να δημιουργήσουμε περισσότερη εμπιστοσύνη. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε συνθήκες εμπιστοσύνη στην αγορά. Θα πρέπει να καταφέρουμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων και εν γέννη νομίζω θα, κατα... θα πρέπει να καταφέρουμε να ανακτήσουμε την διεθνή εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ω θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοβούλιο, Επιτροπή, Συμβούλιο αλλά και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έχουμε έναν κοινό στόχο. Ο καθένα μα στα πλαίσια τη αρμοδιότητά του θα πρέπει να συμβάλλει στο να στεφθεί με επιτυχία το νέο αυτό σχέδιο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ο καθένα θα πρέπει να λάβει προφανώ τι ευθύνε του. Και τώρα ο κύριο Μπούλμαν και μετά όλου οι Κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε για λόγους ε, χρόνου στο Στρασβούργο στις τελικές μου παρατηρήσεις μίλησα μόνο προς την Κομισιόν και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Σήμερα θέλω να στραφώ προς τους συναδέλφους γιατί κάναμε μια συζήτηση επί των τροπολογιών και θέλω σήμερα να αξιοποιήσω το χρόνο για να απαντήσω στους συναδέλφους. Μία προκατακτική γενική παρατήρηση. Βεβαίως, βεβαίως, πάντα έχουμε πίεση χρόνου και ακούσαμε τόση ώρα. Πρέπει και εμεί να μπορούμε να πούμε κάτι. Μία παρατήρηση λοιπόν. Από ό,τι γνωρίζω τις ευρωπαϊκές συνθήκες, η Κομισιόν κάνει νομοθετική πρόταση και μετά το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εδώ πρέπει να συμφωνήσουν επί του νομοθετήματος. Νομίζω ότι εξακολουθεί να ισχύει αυτό. Αντίστροφο ε, συμπέρασμα, η Κομισιόν δεν μπορεί να αποφασίσει μόνη της ε, τα νομοθετήματα. Μπορεί μερικοί να το θέλουν, αλλά εξακολουθούμε να είμαστε στην ε, ενωσιακή νομοθετική διαδικασία. Έτσι πρέπει να γίνουν αυτά τα πράγματα. Το Κοινοβούλιο θα κάνει ό,τι μπορεί, ούτω ώστε σύντομα να καταλήξουμε. Αυτό ισχύει και για την ΕΤΕ. Η ΕΤΕ είναι ε, σε πολύ κεντρική θέση. Το θέλουμε αυτό. Αλλά η ΕΤΕ είναι ένα όργανο της ευρωπαϊκής πολιτικής. Η ΕΤΕ δεν είναι νομοθέτης. Και αυτό είναι σημαντικό να το καταλάβουμε. Γιατί εμείς φυσικά ως Κοινοβούλιο Θέλουμε, θέλουμε να αναλάβουμε πλήρως αξιότιμοι πρόεδροι ε, τις ευθύνες μας. Και εφόσον το καταλαβαίνουμε αυτό, τότε έχουμε από το Συμβούλιο την ευθύνη για να δοθούν αυτές οι εγγύησεις και πρέπει να δώσουμε απαντήσεις. Σεβόμενοι πλήρως την εντολή μας, την εντολή που έχει ο κάθε συνάδελφος. Και οπότε πρέπει να πω ότι με εντυπωσίασε η συζήτηση σήμερα. Διότι σχεδόν ποτέ δεν είναι ένα τόσο περίπλοκο θέμα, ένα τόσο σημαντικό εγχείρημα, όπου ε, συμμετέχουν τόσες πολλές επιτροπές να αντιμετωπίζεται με τόσο ευρεία συνένεση. Τόσο ευρεία συνένεση. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά πολύ κοντά ο στον άλλον και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να καταλήξει σύντομα. Να αναφέρω μόνο μερικά σημεία. Γιατί έχουν ουσιώδη σημασία για να συνεννοηθούμε. Ορισμένοι συνάδελφοι από διάφορε ομάδε, δικαίω, νομίζω, δικαίως νομίζω ανέφεραν ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει το ταμείο αυτό τη διαθροτική μας πολιτική. Και αυτή είναι η πρόθεση και της Κομισιόν. Αυτό το στρατηγικό ταμείο είναι ένας πυλώνας. Άλλοι πυλώνες ε, πρέπει να προωθήσουν διαθροτικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά θέλω να σας καθησυχάσω αγαπητοί συνάδελφοι. Εάν θα μπορούσα μέσω αυτού του εγχειρήματο να διασφαλίσουμε ότι τα χρήματα που δεν αξιοποιούνται θα αξιοποιηθούν εκεί που χρειάζονται, αυτό θα ήταν μια τρομερή διαθροτική μεταρρύθμιση. Πρέπει να είμαστε υπέρ. Κάτι άλλο. Να υπενθυμίσω ένα παράδειγμα που μας ενέπνευσε ιδιαίτερα στα πλαίσια της ακρόασης που κάναμε. Κάποιος κύριος από μια πλατφόρμα έρευνας είχε προσκληθεί από πλευρά των συναδέλφων του ΕΛΚ και μας ε, διηγήθηκε τι υψηλού επίπεδου εμβόλια προσπαθούν να αναπτύξουν και παράλληλα προσπαθούν να δουν τι μπορούν να κάνουν για να ε, μπορέσουν να μειώσουν όλες τις ε, κανονιστικές ρυθμίσεις για να μπορέσουν να τα φέρουν στην αγορά των δυνατών πιο σύντομα. Νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή προσέγγιση των διαθροτικών μεταρρυθμίσεων που χρειαζόμαστε. Υπάρχουν και πολλά άλλα που συζητήσαμε, αλλά είναι κυρίως τεχνικής φύσης και θα βρούμε τις κατάλληλες απαντήσεις. Είμαι απόλυτα πεπισμένος. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους για τη συμβολή τους. Το τελευταίο που θέλω να πω είναι αυτό που είπε ο κύριος Κάρας. Ναι, το θέλουμε και το ταμείο και το χρονοδιάγραμμα. Δεν θέλουμε να αποτύχουμε. Θέλουμε ένα αποτέλεσμα που να μην είναι ετέσιν, να είναι πραγματικά κάτι καινούριο, όπου ο καθένας να μπορεί να συμβάλλει για να ε, επιτύχουμε το καλύτερο για τους ε, συμπολίτες μας. Πρόεδρος, ο κύριος Φερνάνδης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά το ζήτημα της χρηματοδότησης, την πιο δύσκολη αν θέλετε ερώτηση. Εμείς προτείναμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον όρο αμετάκλητη. Εμείς είπαμε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις για την εγγύηση. Θέλουμε και υπερασπιζόμαστε την αξιοπιστία λοιπόν. Και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θέσουμε να αμφιβόλο αυτή την αξιοπιστία. Πρέπει όμως να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί αν έρθει κάποιος και μας πει ότι η δική μας η τοποθέτηση μπορεί ενδεχομένω να οδηγήσει σε μείωση της αξιοπιστίας, τότε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί τότε ενδεχομένω η ίδια η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να είναι εκείνη η οποία θα μπορούσε να φοβήσει, θα μπορούσε να δημιουργήσει μείωση της αξιοπιστίας. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το μόνο το οποίο κάνει είναι ότι μειώνει τις δεσμεύσεις. 3,3 για τον οριζόντα 2020, 2,7 όσον αφορά το, το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη. Στη συνέχεια, σε κάθε χρόνο, θα κάθε χρόνο θα πρέπει να, να χρηματοδοτούμε το Ταμείο Εγγύησης. Κάθε χρόνο θα πρέπει βάση του δημοσιονομικού δελτίου να μπορούμε να δούμε ακριβώς ποια είναι τα χρήματα τα οποία θα βάζουμε σε αυτό το ταμείο και θα πρέπει να γνωρίζουμε τελικά ποια θα είναι η τελική μας η θέση αν τελικά σε ετήσια βάση θα συστήσουμε αυτό το ταμείο εγγυήσεων και θα πρέπει να δούμε αν στο δημοσιονομικό μας δελτίο θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αλλαγές. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι καταστροφική, γιατί και εμείς η τελευταία ανάλυση σε τήσια βάση, χρησιμοποιώντας τα μέσα ευελιξίας, μπορούμε να ξεκινήσουμε με μία αύξηση 10%, να προχωρήσουμε σε μία κάποια μείωση στη συνέχεια κάποιων προγραμμάτων. Έχουμε δηλαδή και εμεί ένα περιθώριο ευελιξίας και βέβαια μετά από συμφωνία με το Συμβούλιο. Συνεπώς, αν πούμε ότι η δική μας η πρόταση ενδεχομένω να θέσει εν κινδύνο στη συνθήκη, αυτό από μόνο του είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί ενδεχομένω αυτό σημαίνει ότι και η ίδια η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει έναν κινδύνο τι συνθήκε. Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε αυτά τα δύο δισεκατομμύρια τη ευελιξία, τα οποία δεν τα εντοπίσουμε πουθενά στον κανονισμό. Και αυτό και πρέπει να το πούμε, διότι ε, δεν μπορούμε εμείς ως ε, συνομοθέτες, ως νομοθέτες να πούμε στην ε, αρμόδια εκτελεστική αρχή για το πώς θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τα μέσα αυτά, ακόμα και το μέσο ευελιξία. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε το Ταμείο αυτό, θέλουμε το Ταμείο να αρχίσει να λειτουργεί τον Ιούνιο, θέλουμε το Ταμείο αυτό να είναι αξιόπιστο, προκειμένου να στεφθεί τελικά με επιτυχία το όλο εγχείρημα. Και έχω, νομίζω, όλοι μας έναν κοινό στόχο. Όλοι μας θέλουμε στο τέλος να καταφέρουμε να μειώσουμε τον αντίκτυπο, τον αρνητικό αντίκτυπο όσον αφορά τις μειώσεις που θα προκύψουν από τον ορίζοντα 2020 και από το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη. Και θα πρέπει το Ταμείο Εγγυήσεων όχι μόνο να ισχύει για το 2014-2015, αλλά και για την, για, για την περίοδο 2014-2020, αλλά και για την περίοδο μετά το 2020. Και αυτό γιατί το Ταμείο Εγγυήσεων θα πρέπει να υπερβεί την περίοδο αυτή, θα πρέπει να υπερβεί το 2020. Δεν θα το χρειαστούμε το Ταμείο αυτό κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων. Μπορούμε πάντως να μειώσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο. Η ε, αναθεώρηση που θα γίνει για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2017 ενδεχομένως να μας δώσει τη δυνατότητα να μειώσουμε τον αρνητικό αντίκτυπο που υπάρχει για τον ορίζοντα 2020 και το μηχανισμό συνδέοντας την Ευρώπη. Όλες αυτές οι τροπολογίες οι 2.730 καταδεικνύουν πραγματικά ότι όλοι μας θέλουμε να βελτιώσουμε το κείμενο αυτό. Θέλουμε ένα ταμείο το οποίο να παρουσιάζει μεγαλύτερη δημοκρατική λογοδοσία. Θέλουμε να επιφέρουμε βελτιώσεις ακόμα και στη διατύπωση που χρησιμοποιείται. Θέλουμε ένα ταμείο το οποίο θα αποτελεί μια πραγματική ευκαιρία, θα αποτελεί μια πραγματική καινοτομία και θα είναι βέβαια και μια νέα πρόκληση. Πρόκληση για τις περιφέρειες, πρόκληση για την έρευνα, πρόκληση για τους πάντες και δεν αναφέραμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Το ότι θα πρέπει να έχουμε και αυτό τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών. Θέλουμε μέσω του κόμβου αυτού, μέσω του κέντρου αυτού να καταφέρουμε να βοηθήσουμε περισσότερο και τις μειονεκτούσες περιφέρειες. Η μη πολιτικοποίηση. Και αυτό το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό θα πρέπει να δούμε πώς θα καταφέρουμε να ενσωματώσουμε αυτή τη μη πολιτικοποίηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Επιτροπή Επενδύσεων, αλλά και στις κατεξουσιοδότηση πράξεις, οι οποίες θα πρέπει να μας απασχολήσουν περαιτέρω. Όσον αφορά την αρχή της προσθετικότητας τώρα, Θέλουμε προφανώς το Ταμείο αυτό, ακριβώς επειδή έρχεται να συμπληρώσει τις υφιστάμενες δράσεις, χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις, χρειαζόμαστε οικονομική ανάκαμψη και γι' αυτό το λόγο θα προχωρήσουμε με το δύσκολο αυτό έργο, ακριβώς επειδή γνωρίζουμε ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες αξίζουν μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία θα έχει οικονομική ανάπτυξη και απασχόληση. Πρέπει λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσωπώντας τους πολίτες αυτούς, να επιτελέσει το ρόλο του. Ευχαριστώ κύριε Σιγητές έχουμε εμπιστοσύνη και τα κράτη-μέλη θα μπορούσαν να δείξουν ότι έχουν εμπιστοσύνη αποδεχόμενα ότι τα πλεονάσματα στο τέλος κάθε οικονομικού έτους θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη χρηματοδότηση του χρηματοδοτικού αυτού ταμείου. Ο κύριος Γκουαλτιέρη. Ναι, ήταν νομίζω πολύ χρήσιμη και επικοδομητική συνεδρίαση. Εκτός από κάποιες παρεμβάσεις που πρέπει να πω ειλικρινά δεν θεωρώ ιδιαίτερα λογικές και επικοδομητικές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρότεινα να αποφεύγονται κάποιες υπερβολικά δημιουργικές ερμηνείες του άρθρου 310 της συνθήκης. Ξέρουμε πολύ καλά τι λέει και τι εννοεί. Παρ' όλα αυτά, βλέπω ότι έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, συγκλίνουσες προσπάθειες από τους συναδέλφους για να έχουμε μια ε, στεναρή και βιώσιμη και έγκαιρη λύση για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα Juncker. Πολύ ενθαρρυντικό είναι το ότι όλες οι παρεμβάσεις δείχνουν ότι πρέπει και από τεχνική και τεχνοοικονομική προσπάθεια πρέπει το πρόγραμμα να είναι ρωμαλαίο και να είναι νέες επενδύσεις αυτές που θα γίνουν. Και αυτό να συνδυάζεται, όπως είπε ο κύριος με τα άλλα κριτήρια και για την πολιτικοποίηση Ελπίζω ότι αυτό που εννοεί η Επιτροπή δεν είναι, για παράδειγμα, ότι τα μέλη του μηχανισμού για την εξυγίανση των τραπεζών είναι πολιτικοποιημένα. Πρόκειται για ανθρώπους που ε, εξηγαίνουν τράπεζες. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως είναι πολιτικοποιημένες αποφάσεις τους. Ελπίζω να συμφωνεί η Κομισιόν. Για το θέμα αυτό το Κοινοβούλιο είναι απόλυτα σαφές. Και θα πρόσθετα ακόμη για τις κατεξοδότηση πράξεις εξοδοτούμε την Κομισιόν, αντί εμεί να βάλουμε τίποτα στον κανονισμό. Αυτό είναι ακριβώ ο τρόπο να αποφύγουμε την πολιτικοποίηση. Η γραμμή μα λοιπόν είναι ακριβώ αυτή. Σεβόμεθα τον διαχωρισμό των εξουσιών μεταξύ νομοθετική και εκτελεστική. Σα εκχωρούμε πολλέ τις αρμοδιότητες αντί να τι βάλουμε στον κανονισμό. Γιατί θέλουμε να αποφύγουμε την πολιτικοποίηση. Εν πάση περιπτώσει, οι συγητές με βάση αυτή τη συζήτηση μπορούν να προχωρήσουν πολύ καλά και είμαι πλήρως πισμένος ότι θα έχουμε ένα πολύ αποτελεσματικό πρόγραμμα Juncker αρχές του δευτέρου εξαμήνου. Συμφωνώ με τα όσα είπε μόλις τώρα ο Ρομπέρτο Γκουαλτιέρη Όντως ήταν πολύ πλούσια η συζήτηση που είχαμε και καταδεικνύει τελικά ότι είμαστε σε θέση να καταλήξουμε στο κείμενο, το επιθυμητό κείμενο, το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων να αρχίσει να λειτουργεί ήδη από το φθινόπωρο του 2015. Και το ζήτημα της εμπιστοσύνης είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να κάνουμε νομίζω μία έκκληση στα κράτη-μέλη να μας δώσουν την απαραίτητη ευελιξία όσον αφορά τα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε στα πλαίσια αυτού του Ταμείου. Και νομίζω ότι ήδη στα τέλη του έτου θα πρέπει να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πλεόνασμα. Άλλωστε κάθε χρόνο προκύπτει πλεόνασμα. Α χρησιμοποιήσουμε λοιπόν στα τέλη του έτου, α μα επιτρέψουν τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουμε το πλεόνασμα το οποίο θα προκύψει. Ήδη από σήμερα το απόγευμα οι σκιώδεις συγητές θα συναντηθούν με τους συγητές για να προσπαθήσουν να καταλήξουν στις συμβαστικές τροπολογίες. Στη μία μισή το απόγευμα θα γίνει αυτό. Η επόμενη τώρα συνεδρίαση, η κοινή μάλλον συνεδρίασή μας, Έκον και Μπάτζ, θα λάβει χώρα στις 20 Απριλίου. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας. Και ας έχουμε αυτοπεποίθηση. Θα τα καταφέρουμε θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα κείμενο αποτελεσματικό. Σας ευχαριστώ πολύ. Λύε τη συνεδρίαση.